yeah. Right, Gazine's back. Okay, I'll start anyway and Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και πριν σας παρουσιάσω τον ε, Γεώργ, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την παρουσία τους στην ακρόαση με την Επιτροπή Ήτρε. Φανήκατε πολύ εγκρατή και πειθαρχημένοι, ιδίω όταν σα ζήτησαν να τοποθετηθείτε για ένα λεπτό. Και είχαμε ήδη αργήσει 20 λεπτά, διότι το τμήμα που αντιστοιχούσε στην Επιτροπή Ήτρε ήδη δεν έγινε σεβαστό. Καλό ήταν λοιπόν να τηρήσουμε λίγο πολύ έστω και χοντρικά το χρονοδιάγραμμα. Σα ευχαριστώ για αυτό. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων για τα λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου με τον φίλο μα τον παλιό μα φίλο, τον ε, δόκτωρα Γερζεμπόφσκι. Για να το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί βουλευτέ, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πάντοτε αισθάνομαι σε στο σπίτι μου και σα έχω φέρει και ένα καινούριο έγγραφο. Ελπίζω ότι το λάβατε. Ιδάλω θα σα μοιραστεί αμέσω. Είναι μια επικυροποιημένη εκδοχή της έκθεσης πρόοδου έξι μήνες μετά την περασμένη μου παρουσίαση. Να ξεκινήσω με τα θετικά στοιχεία. Από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, η Βουλγαρία και η Ρουμανία υπέγραψε μια κρατική συμφωνία για τον Δούναβη στις 20 Δεκεμβρίου πέρσι. Πήγα στη Σόφια και τον Βουκουρέστι και μπορώ να σας πω ότι συνεργαζόμαστε στενά για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη υλοποίηση και για συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και τους ε, παρόχους, τους παρέχοντας τις υπηρεσίες σε σχέση με τα FAB. Νομίζω λοιπόν ότι το τμήμα αυτό του Δούναβη, το λειτουργικό αυτό τμήμα ενέργειου χώρου, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Η Δανία, η Σουηδία Βρετανία και Ιρλανδία μας απομένουν ακόμη να ολοκληρωθούν. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο και ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι για το δανέζικο, βρετανικό, σουηδικό και ιρλανδέζικο ε, τμήμα ε, έχουν εντατικοποιηθεί εργασίες από τους υπεύθυνους φορείς, ενδεχομένως για να υπάρχει και συγχώνευση των FAB αυτών. Λέγεται FAB 4. Δεν είναι τέσσερα διαφορετικά ε, το τέταρτο υπαριθμόν, αλλά είναι το FAB 4 διαφορετικών χωρών. Εδώ λοιπόν, εδώ θέλουμε να δούμε τους φορείς και τη δυνατότητα συγχώνευσης δύο FAB διαφορετικών κρατών σε επίπεδο ευρωπαϊκών φορέων και παρόχων υπηρεσιών και εθνικών. Νομίζω ότι όλη αυτή η πρωτοβουλία είναι θετική. Γιατί και εσεί είχατε παρουσιάσει ένα επιχείρημα στην αρχή τη χρονιά όταν υποβάλλατε έκθεση και την αποστήλατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητήσατε στην ερχόμενη διετία να μειωθεί ο αριθμό των ΦΑΜΠ από 9 σε έναν χαμηλότερο αριθμό, ώστε να οδεύσουμε και προ τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Νομίζω λοιπόν ότι από αυτήν την έννοια το σουηδικό, δανέζικο, βρετανικό και ιρλανδικό Φαμπ, εφόσον γίνει ενιαίο, θα είναι ένα καλό παράδειγμα. Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο πιο στενάχωρες παρατηρήσεις. Πρώτον, τέσσερα θαμπ δεν είναι ακόμη αντικείμενο καν κρατική συμφωνίας. Ξέρετε ότι για να είναι λειτουργικά τα θαμπ πρέπει να υπάρχει κρατική συμφωνία και μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών. Ακόμη και συμφωνία πραγματικής συνεργασίας και ολοκληρωσής επίπεδο εθνικών παρόχων. Έχουμε λοιπόν τέσσερα ΦΑΜ που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο κρατική συμφωνία. Το Βόρειο Ευρωπαϊκό ΦΑΜ, Νορβηγία, Φινλανδία, Εστονία και Λετωνία δηλαδή. Και μπορώ να έχω λίγο καφέ. Και μετά το ΦΑΜ της Βαλτικής, Πολωνία, Λιθουανία. Το τρίτο είναι το νοτιοδυτικό, Πορτογαλία και Ισπανία. Και το τέταρτο αυτό που ονομάζουμε γαλάζια Μεσόγειο, Blue Med, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρος. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα επικοινώνησα με Κυπρίους υπευθύνου και μα είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είπα εγώ. Ε, κυβέρνηση δεν έχουν, θα αποφασίσει ο λαό. Όμω εσεί οι τρει αντωμεταξύ αρχίστε να ετοιμάζετε τα υπόλοιπα. Προετοιμαστείτε λιγάκι. Υπογράψτε κρατική συμφωνία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μετά τις εκλογές στις αρχές Μαΐου στην Ελλάδα θα έπρεξει έστω κυβέρνηση συνασπισμού, οτιδήποτε και αν προκύψει, αλλά κάποιος υπουργό αρμόδιος για τα θέματα αυτά που να αποφασίσει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο απογοητευτικό στοιχείο. Τέσσερα ΘΑΠ δεν έχουν αποτελέσει καν αντικείμενο κρατική συμφωνία. Αλλά κάτι άλλο που είναι πολύ δυσάρεστο είναι ότι έχουμε δύο Θάμπ λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου που έχουν αποτελέσει αντικείμενο κρατική συμφωνία, αλλά δεν έχει υπάρξει πραγματική υλοποίηση, εντατικοποίηση δηλαδή τη συνεργασία. Εάν θυμάστε το ΦΑΝΤΕΚ, το διαβόητο ενίο ευρωπαϊκό ΦΑΜ, 55% του ενέργειου χώρου και 6 χώρε, έγινε αντικείμενο συμφωνία το 2010 ήδη. Όμως ε, έχω θυμώσει. Δεν ε, έχουν εγκρίνει τίποτα ένα χρόνο αργότερα. Σε επίπεδο όμω ε, εθνικών φορέων και εποπτικών αρχών, επίση η πρόοδο είναι ισχνή. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μάλλον τι γαλλικέ εκλογέ. Να δούμε αν έστω η νέα γαλλική κυβέρνηση να λάβει κάποια πρωτοβουλία. Αλλά τελικά δεν μπορούμε να περιμένουμε στην Ευρώπη όλο και τι επόμενε εκλογέ. Και το άλλο φάμπ είναι το φάμπ τη Κεντρική Ευρώπη, FAB το οποίο καλύπτει 7 χώρε θα θυμάστε Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία και Βοσνία Ζεργοβίνη. Και εκείνοι προσπαθούν να βρουν κάποια μέθοδο, αλλά να σας πω την αλήθεια, επισκέφτηκα πρόσφατα τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, γιατί έχουν την Προεδρία του Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και για το FAB-EC και για το FAB-C, το προηγούμενο δηλαδή και αυτό που αναφέρω τώρα, ε, είναι δυσάρεστα τα στοιχεία. Διότι η λογική της νομοθεσίας του S2 ήταν ότι μετά από δύο χρόνια, δηλαδή από το 2009 που εγκρίθηκε, ότι μετά από τρία το αργότερο, 4 Δεκεμβρίου 2012, θα υπάρξει σαφής πρόοδος πλέον ή τουλάχιστον οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δούμε σαφείς βελτιώσεις στα τέσσερα σημαντικότερα ζητήματα. Ασφάλεια, δυνατότητες, αποτελεσματικότητα προ το κόστος και τον αντίκτυπο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ήδη σε κάποια θα είχαμε θετικές ε, επιπτώσεις και να πω ότι δεν είναι το θέμα μας η πλήρης απουσία μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στους τρεις τομείς, ε, με διαφορές βέβαια από FAB σε FAB, όπως η νέα ευθυγράμμιση των αεροδιαδρόμων που πηγαίνει καλά στα περισσότερα από τα Δεν ε, χρειάζεται πλέον κανείς να κάνει τις ίδιες αποστάσεις που έκανε προηγουμένως. Επίσης ε, υπάρχει εξοικονόμηση καυσίμων, αυτό είναι καλό και για το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ευέλικτη χρήση επίσης του ενέργειου χώρου σε κάποια FAB και αυτό είναι μια από τις επιτυχίες των FAB. Και για πρώτη φορά η πολιτική και η αισθητική αεροπορία αρχίζουν να σκέπτονται πώς μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Στις περισσότερες χώρες, όταν μιλώ σε σμινάρχους, μου λένε ότι δεν έχουν αρκετά κονδύλια ίσως για να αγοράσουν τα απαραίτητα καύσιμα και να πλοηγούν 20 μέρες τη εβδομάδα 20 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα, αυτό του ΦΑΠ της Δανίας Σουηδίας. Εκεί ίδρυσαν μια κεντρική εταιρεία ως παρέχοντα υπηρεσίες για την παροχή δηλαδή των υπηρεσιών και θα ξεκινήσει να παρέχει τις υπηρεσίες τη από τον Ιούλιο. Ενιαίος φορέας παροχή υπηρεσιών λοιπόν και εφόσον λειτουργήσει αυτό το, αυτό το παράδειγμα, αυτό το μοντέλο και εφόσον τελικά λειτουργήσει μεταξύ δύο χωρών θα μπορούσε κανείς μακροπρόθεσμα να καταργήσει όλες τις εθνικές αερογραμμές και να λειτουργήσει με ένα κεντρικό φορέα. Έτσι λοιπόν, παρά τι αποκριτικέ παρατηρήσει και το πώ έχουν προχωρήσει τα πράγματα και από τα ΘΑΜΠ, η ουσία είναι ότι για κάποια από αυτά υπάρχουν θετικά βήματα πρόοδου. Έχουν πολλά να προσφέρουν στου πολίτε μα. Μιλάμε για ένα εργαλείο που μπορεί να μα επιτρέψει να πετύχουμε πραγματική πρόοδο για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Επίση, έχουμε και ένα άλλο εργαλείο. Τα προγράμματα εθνικών επιδόσεων. Εάν θέλετε να διαβάσετε κάτι σχετικά, μην διστάσετε θα δείτε για κάθε φαμπ τουλάχιστον ε, δικές μου παρατηρήσεις ε, σε σχετική έκθεση και την προσωπική μου αποτίμηση για το πώς οι εθνικές προτάσεις σε σχέση με τις επιδόσεις είναι αποτελεσματικές. Εγώ μόνο τέτοιε αποτιμήσει μπορώ να κάνω. Ελπίζω να μην θέλω να με σκοτώσουν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, αλλά έπρεπε να κάνω και προσωπικά σχόλια. Ε, διότι ο φορέα ε, παρακολούθηση των επιδόσεων. Αυτή τη στιγμή περατώνει το έργο τότε Την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιευτεί η σχετική έκθεση και θα τα δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, είναι δική μου προσωπική τελείωση αποτίμηση. Αλλά εάν δείτε ότι στο καλό ΦΑΜΠ του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανία σχολιάζω ότι η Βρετανική και Ιρλανδική αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τι επιδόσει είναι συμβατή με του ευρωπαϊκού στόχου, αλλά με την παρατηρήση ότι η Μεγάλη Βρετανία ζητήθηκε του στόχου περικοπή του κόστου να του αναθεωρήσει. Χωρί αρκετέ ε, ικανοποιητικέ αλλαγέ όμω. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε το μήνυμα, αλλά περί επιδόσεων και των προγραμμάτων τους η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει μόνο δις από τα κάτι μέλη. Βελτιώστε τους στόχους σας βελτιώσετε τι επιδόσει Αλλά δεν έχει δυνατότητα να του προσάγει. Στην περίπτωση. Συνήθω. Αλλά στην περίπτωση των ΦΑΠ, τα κράτη-μέλη μπορούν να προσαχθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφόσον δεν υλοποιήσουν τα των ΦΑΠ εγκαίρω και επί τη ουσία. Να πω, ολοκληρώνοντα, ότι νομίζω καλό είναι να θυμηθούμε στα κράτη-μέλη ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη, ομοφόνος μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο, συμφώνησαν αυτή την νομοθεσία. Άρα έχουν την αρμοδιότητα να την υλοποιήσουν. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να τα φροντίσουν, να τα οργανώσουν σωστά τα φάμπ και μάλιστα εγκαίρως. Έχουμε κάποια καλά παραδείγματα. Εάν λοιπόν κάποια μέλη είναι αποτελεσματικά δεν καταλαβαίνουμε γιατί τόσο πολύ δυσκολεύονται άλλοι το εξηγούμε. Τι έκαναν οι άλλοι αποτελεσματικά για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερε δυνατότητε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προ το κόστο και λιγότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Άρα λοιπόν να θυμηθούν τα κάτι μελη ότι πρέπει να βιαστούν. Να βιαστούν για να ολοκληρωθεί η δουλειά του ω τι 4 Δεκεμβρίου. Και εσεί θα μπορούσατε να μιλήσετε στου υπουργού μεταφορών σα σε εθνικό επίπεδο και να του πείτε, να τους πείτε αυτό ο τραγικό ε, συντονιστή των ΦΑΜΠ έχει κάνει φρικτέ παρατηρήσει στην εκθέση του. Κάνε κάτι. Προσπαθείτε να, προσπαθήστε να τους πιέσετε. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν. Όλοι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη ώστε να φτάσουν στον επιδιωκόμενο στόχο. Σας ε, βεβαιώ ότι ο αντιπρόεδρος Κάλλας που μόλις χθε τον συνάντησα βλέπει τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό ως μία από τις βασικές του αρμοδιότητες για το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς. Γνωρίζει επακριβώς ότι το Κοινοβούλιο περιμένει να δει τι κάνει. Η Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακα των συνθήκων. Εάν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τη δουλειά του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να του στείλει επιστολέ προειδοποιητικέ. Και εγώ το πρότεινα αυτό. Είναι σαν μια προετοιμασία για διαδικασία του παραβάση. Ο χρόνο περνάει τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στις 5 Δεκεμβρίου φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αρχίσει να στέλνει ε, τις επιστολές και τη διαδικασία επιπαραβάσεως. Μην απατώμεθα την προσπάθεια αυτή για τον ευρωπαϊκό ουρανό. Την αναλάβαμε υποσχόμενοι στους πολίτες ότι ο ουρανός αυτός θα δημιουργηθεί, ότι θα είναι θετικές οι συνέπειες για τους πολίτες, τον οικονομία και το περιβάλλον. Μην το ξεχνάμε. Εμείς το εννοούσαμε αυτό όταν δεσμευτήκαμε. Το λέω και ενώπιον του Κοινοβουλίου. Άλλωστε, α αναρτηθούμε. Πόσο συχνά έχουμε σχεδιάσει ωραιότατε νομοθεσίε και τελικά δεν τι έχουν μεταφέρει τα κράτη-μέλη ποτέ. Είναι λοιπόν θεματοφύλακα εδώ η Επιτροπή και ακριβώ ο ρόλο μα είναι να εγκαλέσουμε όλου την τάξη. Έτσι του βλέπει τουλάχιστον ο κύριο Κάλλα. Ξεκίνησα με τι θετικέ παρατηρήσει. Θέλω να κλείσω λοιπόν και μια, μια θετική παρατήρηση. Ήδη τρίτε χώρε μιλάνε για προσχώρηση στα ΦΑΜ. Ξέρετε ότι βάσει τη νομοθεσία ε, ο στόχο των ΦΑΜ. Μάλλον η λειτουργία των ΦΑΜ είναι εντό τη αρμοδιότητα των 100 μελών. Δεν μπορεί η Επιτροπή να παρέμβει και να του πει πώ να συνεργαστούν με άλλου. Τα κράτη-μέλη μπορούν να καλέσουν τρίτα κράτη να συμμετάσχουν. Ωραία θα ήταν λοιπόν ενδεχομένω να μιλήσουμε και με άλλου και να δούμε τι ιδέε έχουν. Η Ισλανδία ήδη έχει κάνει κρούση. Ο υπουργό ε, που είναι υπεύθυνο για τι μεταφορέ ε, επικοινώνησε μαζί μου και νομίζω ότι θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά σε ποιο θα μπορεί να συμμετάσχει και υπό ποιε προποθέσει. Ήδη συμμετείχε στην πρώτη φάση του NE Έφυγαν από εκείνη την ομάδα, αλλά θα μπορούσαν να επιστρέψουν. Σκέφτηκαν το σουηδικό-δανέζικο φαμπ, διότι η Ισλανδική αρχή συμφωνεί με την ε, κυβέρνηση της Δανίας ώστε να εκμεταλλευτούν το κοινό τους έργο για την Γρινλανδία και τις ε, σχετικές ε, μεταβιβάσεις και επίσης υπάρχει σχέση και με το Βρετανικό Ιρλανδικό Φαμπ και ως προς τις συλλογή εσόδων από την αρχή. Αλλά αν δείτε και τους αεροδιαδρόμους από το βορρά περνάνε από την Ιρλανδία και τη Βρετανία. Η Ισλανδική λοιπόν κυβέρνηση έχει επιλογή μεταξύ τριών φαμπ στην ουσία. Όμως θα δουν από ποιον πρέπει να προσκληθούν και κατά πόσον θα προσκληθούν. Και εγώ έχω επιστήσει την προσοχή των ε, ευρωπαϊκών κρατών σε αυτόν τον τομέα. Κάτι άλλο, ε, πήγα και στη Σερβία Εάν δείτε στην πρώτη μου σελίδα, το αναφέρω εδώ, υπάρχει ένα κενό εδώ μεταξύ του ΘΑΠ του ΘΑΠ του Δούναβη και της ε, Μεσογείου. Εδώ λοιπόν, ε, μεταξύ αυτών των τριών χωρών, κάποιες έχουν καθεστώς υποψήφιων για προσχώρηση. Η Βοσνία, Ριζεγοβίνη και η, η Σερβία. Η Σερβία λοιπόν, όπως έλεγα, έχει ουσιαστικά μια εσωτερική συμφωνία θα, με το Μαυροβούνιο, και έχει και αρμόδια αρχή ε, που αναλαμβάνει την ε, επικοινωνία μεταξύ Σερβία και Μαυροβουνίου. Εδώ οι εξελίξει ω τώρα ήταν θετικέ Συνομίλησα και με τους Ρουμάνου και Βουλγάρους, μέλη του ΦΑΜΠ του Δούναβη, και θα δούμε ποιον θα προσκαλέσουν. Αλλά αν το δείτε από μια άλλη πρόπτικη, ε, καλή δεν θα ήταν και η Μολδαβία να τοποποιήσει τις συζητήσει τη με την Ρουμανία και Βουλγαρία. Από τα ανατολικά ίσω. Από την άλλη θα μπορούσε να συμμετάσχει και από τα δυτικά. Η Σερβία λοιπόν και το Μαυροβούνιο, εφόσον έχουν ήδη κρατική συμφωνία, καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν. Ενδεχομένω και η Μακεδονία, η οποία επισήμω ονομάζεται Φύρομ, τέλο πάντων Μακεδονία. Η Μακεδονία λοιπόν θα μπορούσε και αυτή να προσχωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν ποιο να προσκαλέσουν ε, στα ΘΑΜ. Όμω θεωρώ, βήμα. Μάλλον θεωρώ ότι είναι θετικό βήμα οι χώρες αυτές, ε, ότι οι χώρε αυτέ μπορεί να προσκληθούν και κάποιε άλλε από τα Δυτικά Βαλκάνια σκέπτονται την προσχώρησή του στο σύστημα των ΘΑΜ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θετικά όλα αυτά τα στοιχεία και ολοκληρώνοντα να σα πω ότι η Γενική Διεύθυνση Μούβ με το προσωπικό τη μα εξυπηρέτησε ιδιαίτερω. Του βλέπετε στο πίσω μέρο τη αίθουσα, ο κύριο Μπόλτουεν, ο διευθυντή, ο υπεύθυνο υπηρεσία, ο κύριο Καστιλέτη και ο κύριο ο οποίο είναι άμεσος συνεργάτης μου, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το έργο, αλλά είναι πραγματικά διασκεδαστικό και χρήσιμο. Γνωρίζετε ότι συχνά τα κάτι μέλη έχουν επίγνωση των υποχρεώσεών τους, αλλά οι Υπουργοί Μεταφορών έχουν προβλήματα με του σιδηροδρόμους, με τα φορτηγά και άμα δεν πέσει και κανένα αεροπλάνο, θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά. Δεν ασχολούνται και πολύ με την αεροπλοεία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να θυμίσουμε σε κάποιου από του μεταφορών ότι υποσχέθηκαν να έχουμε αποτελεσματικότερο ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Δεν τον κάνουμε για την πλάκα μα αυτό. Δεν τα δημιουργούμε τα θάπια σκοπού ε, πνευματική ιδιοκτησία. Θέλουμε να αποκομίσουμε κέρδη στην ασφάλεια, την ε, αποτελεσματικότητα προ το κόστο, τι δυνατότητε και τον περιβαλλοντικό, αντίκτυπο. Αυτό είναι ο στόχο. Όφελο για του πολίτε και για εμά του ίδιου. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαζεμπόφσκι. Οχτώ μιλητέ έχω στον κατάλογο, για... έχουμε 35 λεπτά στη διάθεσή μα και σα παρακαλούσα θερμά να είστε σύντομοι, Δύο μισή με τρία λεπτά το πολύ μπορούμε να προσθέσουμε και τον κύριο Baldwin και να απαντήσει ο George. Αρχίζω με τον κύριο Γκρός. Σε ευχαριστώ Γκέορκ, σε ευχαριστώ Πρόεδρε, σε ευχαριστώ ε, για την θαυμάσια εργασία την οποία έκανες Γκέορκ εθελοντικά μάλιστα, ε, αλλά ε, το αποτέλεσμα είναι λίγαν απογοητευτικό. Και είναι απογοητευτικό διότι όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση. Το Συμβούλιο Υπουργών αποφασίζει και δεν εκτελεί. Εγώ λοιπόν ως απλός πολίτης πώς μπορώ να εξηγήσω σε έναν πολίτη της περιφέρειάς μου ότι πρέπει να σέβεται τον νόμο ενώ εμείς που νομοθετούμε δεν δίνουμε το καλό παράδειγμα. Και πολλές φορές εκεί που διακυβεύεται η φήμη της Ευρώπης και εκεί ιδιαίτερα όπου εμείς έχουμε συμφέρον να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή δομή, πρέπει να ζητήσουμε ευθύνη από τα κράτη τα οποία δεν βοηθούν, δεν υποστηρίζουν. Βεβαίως πάντοτε τίθεται το ζήτημα της εξοικονόμησης ε, χρημάτων, εξοικονόμηση κόστους. Τι πρόγραμμα λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής πρέπει να εντοπίσουμε τις δυσκολίες. Ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες τέλος πάντων που εμποδίζουν την εκτέλεση των ε, συμβάσεων. Ποια είναι τα προσκόμματα. Δεύτερον, η εθνική στόχοι. η εθνική στόχοι είναι στη δεύτερη φάση και είναι τμήμα του προγράμματος. Ποια είναι λοιπόν τα προσκόμματα στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων και πώς μπορούμε να τα κάνουμε πιο αποδοτικά. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ερώτημα αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση για τα εικονικά κέντρα, τα virtual centers και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του προγράμματος CESAR για να αναπτυχθούν αυτά τα εικονικά κέντρα και να επιταχύνουν την εξέλιξη των FAB. Εν κατακλείδη θέλω να πω ότι, ότι αναμένουμε μία πολύ σκληρή στάση της Κομισιόν και πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο να περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους να μας ξαναπούνε αυτά τα οποία ήδη ξέρουμε. Έχουμε ήδη στείλει τις ε, επιστολές και θέλουμε να επιταχύνουμε το έργο και από το Δεκέμβριο του 2012 επιτέλους να αρχίσει η υλοποίηση. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τους, συναδέλφους, τους συναδέλφους, τον κύριο Γιαζεμπόφσκι και τον κύριο Γιαζεμπόφσκι για την ειλικρινή ανάλυση της κατάστασης. Δεν είναι ότι απογοητευόμαστε, ξέρουμε πώς τα εφαρμόζουν όλα αυτά τα κράτη-μέλη και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση. Αναφέρατε κι εσείς όλα τα πλεονεκτήματα των FABs και η μεταρρύθμιση είναι γενικά γνωστή. Θα υπάρχει περισσότερη αποτελεσματικότητα, χαμηλότερο κόστος, λιγότερη ρήπανση. Όλα αυτά είναι θετικά βέβαια. Φυσικά χρειάζεται μια στρατηγική έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόζουν όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η καταλληλότερη για να προχωρήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια μπορεί να κάνει πολλά, αλλά ο αντίκτυπος είναι μικρότερος. Άρα βραχυπρόθεσμα τα κράτη-μέλη πρέπει να πιστούν επίσημα να τηρήσουν την προθεσμία. Υπάρχει και ένα δεύτερο βέβαια που πρέπει να σκεφτούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα που είμαστε στην αρχή να προετοιμαστεί αν μη τι άλλο, έτσι παρασκηνιακά και να ετοιμάσει νέα νομοθεσία που επίγει και να είναι έτοιμη γρήγορα ώστε να μας παρουσιαστεί μετά τις προθεσμίες. Κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω κύριε Γερζεμπόφσκι, Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχει τέτοια καθυστέρηση. Γιατί υπάρχει αντίσταση από τις εθνικές αρχές, γιατί περί αυτού πρόκειται, περί κάτι άλλου. Και πέρυσι, στα πλαίσια της επικουρικότητας που στηρίξαμε τα FAPS, εσείς η Επιτροπή φρόντισε να υπάρξει χρηματοδότηση ώστε να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάσινερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Γκέορκ για την ε, παρουσίασή σου. Ε, Ματιέ ήδη, ήδη είπε ότι είναι τρελό να νομοθετούνται θέματα στα οποία συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη και μετά να γυρίζει κανείς στην έδρα του και τίποτα να, να μην γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν και λένε ότι υπάρχουν ορισμένα προσκόμματα και γι' αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά σε αυτό ειδικά το πρόγραμμα δεν τίθεται ζήτημα αριθμών, απλώς ζήτημα συνεννόησης είναι και στη Γερμανία που οι συζητήσεις ε, συνεχίζονται. Δεν έχουμε προχωρήσει ούτε στη Γαλλία ούτε στη Γερμανία. Κάθε χρόνο προβάλλονται νέες δικαιολογίες. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πιέσουμε όλα τα κράτη-μέλη, το καθένα να προχωρήσει ε, στο δρόμο που έχουμε αποφασίσει. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε, διότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευχάριστη, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Και και εγώ πάντοτε μιλάω υπέρ των, ε, του ευρωπαϊκού ουρανού, ενιαίου ουρανού. Ε, ξέρω ότι πολλά θέματα εξελίσσονται, ξέρω ότι είναι ένα θέμα αγαπητό και προσφυλές, αλλά πολλοί βρίσκονται ακόμα στο σκοτάδι. Ε, δεν ξέρουν ότι συμβαίνουν, ότι υπάρχουν και προγράμματα τα οποία εξελίσσονται στον εναέριο χώρο. Όλοι σκέφτονται συνήθως χερσαία προγράμματα, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, οδικά δίκτυα κτλ. Αλλά σας είπα ότι έχουμε εδώ ένα τείχο μπροστά μας ανοησίας, απογοήτευσης ε, και εκνευρισμού. Επιτέλους πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ ο κύριος Κράμερ. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Μία πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία ιδέα, όλοι συμφωνήσαμε ότι θα έχει μεγάλο όφελος, οικονομικό, όφελος στο θέμα της ασφάλειας, γενικά δηλαδή μια ωφέλιμη προσπάθεια. Τώρα, η υλοποίηση. Πάρα πολύ αργή, πολύ, πολύ καθυστερή, πολύ περισσότερο από ό,τι επισημούσα και εν ώψη της οικονομικής κρίσης θα, θα πίστευα ότι θα προχωρούσε γρηγορότερα, ιδίως όσον αφορά και ε, την ομάδα πίεσης που υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος. Πρέπει κάπου να υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να πιέσει, μια ομάδα η οποία να είναι αποτελεσματική και δραστήρια. Η Αυστρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το FAB Κεντρικής Ευρώπης και θέλει να παίξει ένα δημιουργικό ρόλο δεν ε, μου κάνει εντύπωση ότι τα πράγματα προχωράνε με ρυθμό χελώνας, διότι μέχρι πρόσφατα η Κεντρική Ευρώπη ε, είχε κράτη τα οποία ήταν σε εμπόλυμη κατάσταση μεταξύ τους. Εντάξει, πρόσφατα ξεκίνησε αυτό. Έχουμε μία ε, γενιά το πολύ, μία γενιά ελευθερίας και συνεργασίας. Μπορεί και σε αυτό να οφείλεται μια καθυστέρηση. Αυτή είναι μία δικαιολογία, αλλά δεν τα συγχωρώ όλα. Τώρα, δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει το, τα FAB στις, στις άλλες περιοχές, ε, στους άλλους τομείς. Υπάρχει αντίρρηση συνεργασίας, υπάρχουν προσκόμματα ή ε, σκράτη που δεν θέλουν να συνεργαστούν ε, μαζί με άλλα. Δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς η περιοχή της Μεσογείου, το Blue Med Fab. Ρομαντικό όνομα έχει αυτό, η Γαλάζια Μεσόγειος, το ΦΑμπ της Γαλάζιας Μεσογείου. Εδώ θέλω να ρωτήσω εάν έχει λυθεί έστω εν μέρη το πρόβλημα με τον ε, ε, αέριο χώριο της Βόρειας Ιταλίας, όπου εκεί πάντοτε είχαμε προβλήματα. Έχει λυθεί ή όχι. Και όσον αφορά αυτό το ΦΑΜ, το Μεσογειακό σε σχέση με τα άλλα ΦΑμπ πιστεύετε ότι το ΦΑΠ Κεντρικής Ευρώπης λειτουργεί, είναι μάλλον σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τα άλλα, είναι ας πούμε στον πάτο. Γιατί αν πιστεύετε ότι είναι το χειρότερο και το πιο στάσιμο ας πούμε και το πιο καθυστερημένο πρέπει να δούμε μια στρατηγική να το βγάλουμε από αυτή την κατάσταση, να προχωρήσει. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Γκέροκ για την εξαιρετική του παρουσίαση όλοι είμαστε εν γνώση της ε, δύσκολης εργασίας την οποία επιτελεί. Εγώ είμαι Βρετανή και βεβαίως χαίρομαι ιδιαίτερα που η Βρετανία και η Ιρλανδία έχουν προχωρήσει σημαντικά. Ε, όσον αφορά τα υπόλοιπα προβλήματα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθυστέρησης. Ιδίω στις περιπτώσεις που οι χώρες έχουν υπογράψει και έχουν δεσμευθεί ας πούμε να προχωρήσουν το θέμα αυτό και δεν έχει γίνει τίποτα δύο-τρία χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και για να ενημερώσω τον Γκέορ, τον Τζόρτζ, έχω σχεδόν ολοκληρώσει την έκθεση της ΣΕΤΑ και μας, ε, και βλέπουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε τα ΦΑΠ να προχωρήσουν για να προχωρήσουν και όλα τα άλλα θέματα που συνδέονται με τον, ε, με την, ε, με τον Ευρωπαϊκό Ουρανό. Τους Ευρωπαϊκούς Ουρανούς. Πιστεύω λοιπόν ότι κοιτάζοντας την νότιο-δυτική Ευρώπη ε, την μεσογειακή, ε, το μεσογειακό ΦΑΜΠ, εκεί υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα ευέλικτης ε, χρήσης του ενέργειου χώρου. Η νότιο-δυτική Ευρώπη έχει μεγάλα προβλήματα απασχόλησης συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ΣΑΗ. Εάν ας πούμε δεχτούμε ότι η Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο που βρισκόμαστε ας πούμε στην άκρη της Ευρώπης, έτσι δεν είναι. Και ενώ εμείς είχαμε, ήμασταν πάντοτε εξαιρετικά συντηρητικοί όσον αφορά τη διαχείριση των ουρανών και του ενάριου χώρου και της αεροπλοείας. Αν δείτε όμως τώρα, εμείς έχουμε προχωρήσει, έχουμε προοδεύσει σε αυτό τον τομέα, έχουμε συνεργαστεί και επίσης υπάρχουν θαυμάσιες ευκαιρίες ε, απασχόλησης ε, στην Ευρώπη, βελτίωσης της ασφάλειας, ε, εξοικονόμησης πιστώσεων. Λοιπόν, είναι ανόητο να μην προχωράει το θέμα όλοι, όλοι καταλαβαίνουν τα ωφέλη. Αυτοί λοιπόν που δεν συμφωνούν ή τσακώνονται ή δεν μπορούν να συνεργαστούν, ε, βλάπτουν τον εαυτό τους. Πιστεύω ότι έχουμε εξαιρετικούς ε, εμπειρογνώμονες ε, που αμείβονται πάρα πολύ καλά και δεν ανησυχούν καθόλου για την ε, δουλειά τους, οι οποίοι δεν προσφέρουν τις υπηρεσίε που θα έπρεπε για να προχωρήσει το θέμα. Σε ευχαριστώ λοιπόν George και εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειές σου. Εδώ η αιστεία είναι ανοιχτή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πετύχουμε τα γκολ. President. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γιαζεμπόφσκι για την δουλειά που έχει κάνει. Ξέρω ότι εργάζεστε σκληρά, όμως η πραγματικότητα είναι η εξής. Το Δεκέμβριο 2012 έχουμε την προθεσμία που, που λύγει του, τον ΦΑΜ και ούτε ένα δεν θα είναι λειτουργικό. Αυτό είναι σαφέστατο. Έχουμε λοιπόν προχωράμε προς την τελική προθεσμία και τα πράγματα δεν είναι, δεν εξελίσσονται καλά. Εγώ δεν ήμουν εξ αρχής ε, οπαδός ε, του, της ιδέας αυτής των ΦΑΠ, διότι εγώ έλεγα ότι μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην, ε, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό χωρίς τα ΦΑΠ. Πιστεύω ότι δημιουργούν κάποιο, αν θέλετε, στο ψυχολογικό εμπόδιο. Τι θα κάνετε τώρα μέχρι το Δεκέμβρη που θα εκπνεύσει η προθεσμία. Τι πιστεύετε ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει κάτι. Ε, η προσέγγιση που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα δεν δούλεψε. Και πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μία προσέγγιση από ιεραρχική, από ψηλά προς τα κάτω και όχι από τη βάση προς τα πάνω. Αυτή απέτυχε. Τώρα, εφόσον έχουμε πει ότι θα οργανωθούν αυτά τα, τα FABs, καλό είναι να λειτουργήσουν, να, να γίνουν λειτουργικά. Διότι δεν... Το ερώτημά μου είναι λοιπόν τι μπορεί να γίνει, τι θέλετε εσείς να γίνει και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Κομισιόν μέχρι το Δεκέμβριο 2012. Δεύτερον, αυτή η πρωτοβουλία Α6 ξέρετε τι εννοώ το 70% του ε, ε, που είναι το Α6 πρωτοβουλία A6 6 κρατών που προσπαθούν να ενοποιήσουν τον Ευρωπαϊκό Ουρανό μέσω του προγράμματος απόδοσης A6 λέγεται αυτή η πρωτοβουλία, Α6. Εγώ έχω μιλήσει με ορισμένους εκπροσώπους αυτής της πρωτοβουλίας και έχουν, μου είπαν ότι έχουν καλή πρόθεση, ίσως η καλή πρόθεση είναι προσωπικά δική τους και όχι δεν καλύπτει και τις αρμόδιες αρχές των ε, κρατών τους. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς επιδιώκουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ο κύριος Ντανιέλης, τρία λεπτά. Δανέλης. Ζεμπόφσκι για την ενημέρωση και για τη δουλειά που έχει κάνει για όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, έχω δύο-τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη ε, αναφέρθηκε ήδη από το ΣΑΙΔ, ε, αλλά οι πραγματικοί λόγοι που εσείς εκτιμάτε ότι ε, υπάρχει αυτή η στάση από τα κράτη-μέλη είναι λόγοι πολιτικής βούλησης ή είναι λόγοι γραφειοκρατίας, αδράνειας, προσκομμάτων της διοίκησης. Ε, και επίσης είμαι περίεργος ε, αν έχετε εικόνα του ποια είναι η στάση, η άποψη των αερομεταφορέων, δηλαδή των, αεροπορικών εταιριών. Λειτουργούν ή μπορεί να λειτουργήσουν ως ομάδα πίεσης ή ως ομάδα ανάσχεσης. Επίσης, ε, εκτιμάται ότι αν ε, αρχίσουν να κινούνται ε, τα κράτη-μέλη. Ε, ο, ο ορίζοντας χρονικός της 4ης Δεκεμβρίου είναι αντικειμενικό σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση των ΦΑΜΣ. Ε, επίσης θα με ενδιέφερε αν μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα σε περίπτωση που υπάρχει πολιτική βούληση εν τέλει και τα προβλήματα είναι γραφειοκρατικά περισσότερο το να περπατήσουν τα FABs της ε, νότιας ε, ε, Ευρώπης, που δέχονται το, η περιοχή που δέχεται βεβαίως πολύ αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Είναι ρεαλιστικό να ολοκληρώσουν μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια την θεσμοθέτηση και λειτουργία τους. Τέλος, πέρα από τις συνομιλίες μεταξύ των χωρών μελών και την αντιμετώπιση των διαφορετικών κατά περίπτωση προβλημάτων, σε αυτές τις διεργασίες υπάρχει και εμπλοκή της Επιτροπής Ενίου Ευρωπαϊκού Ουρανού που μπορεί να μεταφέρει τις καλές εμπειρίες, τις καλές πρακτικές ουσιαστικά από τον ένα ΦΑΜ που έχει περπατήσει ουσιαστικά του ε, Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Ευχαριστώ. Mr. Kramer, Τρία λεπτά ο κύριος Κράμερ. Χαίρομαι. Ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπω. Σαν το σπίτι σας εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ποια είναι τα αίτια, ποιοι είναι οι λόγοι. Ε, σίγουρα δεν φταίει ο συντονιστή, διότι πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Άρα λοιπόν άλλοι φταίνε. Όπω είπε και ο Ματιό Γκρό, αυτό το φαινόμενο παρα, σημειώνεται ε, και σε άλλου τομεί, Ακόμα και στην ε, συμμόρφωση, στο cross acceptance, ε, πάλι υπάρχουν καθυστερήσεις και προσκόμματα. Ούτε ενιαίο εισιτήριο υπάρχει, ούτε ενιαίο ουρανός. Ε, μα τι γίνεται επιτέλους. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε γρηγορότερα από το σιδηροδρομικό πακέτο. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αν τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει και δεν σέβονται την υπογραφή του, υπάρχουν κυρώσει. Έτσι δεν είναι. Και η πρώτη ζημιά είναι ότι δεν του εμπιστεύονται οι πολίτε. Εάν οι υπεύθυνοι δίνουν στραβό παράδειγμα, απογοητεύουν και τους πολίτες. Σας ρωτώ λοιπόν ε, πώς μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε και από την Κομισιόν τι, στο καλό έχουν κάνει μέχρι τώρα, τι προγραμματίζουν και πότε μπορείτε να μας υποβάλλετε μια έκθεση που θα λέει ότι έχουμε υπευθύνω κάνει το α, το β και το γ. Ευχαριστούμε πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, κύριος Μπόλτουιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιαρζεμπόφσκι για την εξαίρετη παρουσίασή του. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τι απόψεις του και χαιρόμαστε πολύ που συνεργάζεστε τόσο στενά μαζί μας. Επιβεβαιώνω επίσης ότι ο Αντιπρόεδρος όντως δίνει μεγάλη προτεραιότητα στον, ε, στους ευρωπαϊκούς εθέρες και προσπαθούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Οπότε χαίρομαι που και εσείς μας πιέστε να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Να επιβεβαίωσω τώρα κάτι για τις ημερομηνίε. 4 ε, Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία, είναι δύσκολο να το πετύχουμε. Τέσσερα από τα νέα ΦΑΒΣ έδωσαν ε, τα, τις παρουσιάσεις τους, εκθέσεις τους για το πώς έχουν προχωρήσει. Πιέζουμε βέβαια πολύ και θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη προκειμένου να ε, δημοσιευθούν τα φάβζα στην επίσημη εφημερίδα πριν από την 4η Δεκεμβρίου. Όμως ακούω τα σχόλιά σας που λέτε ότι δεν θέλετε να καθίσετε και να περιμένετε την 4η Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή επίσημα δεν μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση παρά μόνο μετά. Καταλαβαίνω βέβαια που λέτε ότι δεν θέλετε να περιμένουμε και να σκεφτούμε την ιδέα αυτή για μια επιστολή προειδοποιητική που προτείνει ο κύριος ε, Γιαζεμπόφσκι. Σίγουρα και ο κύριος ε, Κάλλας θα το σκεφτεί και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακούω επίσης κάποιους από εσά να λένε ότι πρέπει να ετοιμαστεί νέα νομοθεσία πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των όσων ήδη υπάρχουν. Αλλά πράγματι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα φροντίσουμε εφόσον υπάρχει η ανάγκη να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα. Δεν ξέρω κύριε Μπόλτιν πόσο θα τα καταφέρετε, και, αλλά σίγουρα πρέπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνετε ό,τι μπορείτε. Ο κύριος Γιαζεμπόφσκι. Ελπίζω να μην ξεχάσω τις ερωτήσεις κάποιων. Θα προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω τα ερωτήματα. Με ρωτήσατε ποιες είναι οι δυσκολίες. Εξαρτάται από το κάθε FAB. Σε επίπεδο κρατικό. Κύριε Λιχταμπέργκερ. Είναι θέμα ιστορίας Κάποιοι δεν θέλουν να επιστρέψουμε σε κάποιο είδους αυτοκρατορία, imperium. Τέλος πάντων είναι και ιστορικοί λόγοι κάποιες φορές. Όμως η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή τόλμη από την πλευρά των Υπουργών Μεταφορών. Γιατί, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα διότι οι παρόχες αεροπορικών υπηρεσιών είναι πολύ ισχυρά λόμπι σε κάποιες χώρες και οι υπουργοί αδύναμοι. Ως αποτέλεσμα λοιπόν έχουμε ένα μπλοκάρισμα, ενώ θα πρέπει να έχουν μακρόπνοα σχέδια οι υπουργοί, να έχουν την πυγμή και να πούν Ωραία, ξεκινάμε και συνεργαζόμαστε με τους ομολόγους μας εντός του ίδιου ΦΑΜ. Σε κάποια Φαμ πιστεύουν ε, υπάρχει αίσθηση, μάλλον ότι παρασπίζονται τα εισοδήματά τους, τον ενέργειο χώρο τους, ε, το προσωπικό τους, οι εποπτικές αρχές. Η ε, Δανέζικη υπηρεσία λόγου έχει 6.000 προσωπικό. Ξέρω ότι κάνουν 3.000, αλλά ψάχνω πού ακριβώς απασχολούνται οι υπόλοιποι 3.000. Είναι ακόμα μυστήριο για μένα. Λοιπόν, υπάρχει εσωτερική πίεση από τις εσωτερικές υποπτικές αρχές Θέλουμε να κάνουμε αλλαγέ, αλλά ο καθένα θέλει να υπερασπιστεί το έδαφο του και το εισόδημά του. Πιεζόμαστε από τα κράτη-μέλη. Αλλά αν συγχωνεύσουμε τα προσωπικά υπηρεσιών, εάν συγχωνεύσουμε πόρου, μπορεί όλα να είναι αποδοτικότερα, αποτελεσματικότερα για του πολίτε. Και μάλιστα εφόσον συνεργάζονται προ στιγμή, έχουμε πρόβλημα. Μέχρι πέρυσι μπορούσα να πω στι συνδικαλιστικέ οργανώσει ότι Υπάρχουν πρόπτικε απασχόλησης στην αεροπλοεία. Μη φοβάστε αν γίνεται αποδοτικότεροι. Στατιστικώς τουλάχιστον κάποιοι που θα απολυθούν θα είναι χρήσιμοι γιατί μεγαλώνουν οι ανάγκες της αεροπλοείας. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τι έχει γίνει. Σε κάποια μέρη της Ένωσης έχουμε μείωση στις ε, υπηρεσίες αυτές. Όμως δεν μπορεί η αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και οι σχετικές ε, ιδέες που θα έπρεπε να είναι χρήσιμες για τους πολίτες να παραμένουν καινογράμμα. Το πρόβλημα είναι ότι το κόστος των εποπτικών αρχών, το ανακτούμε, επιστρέφεται από τις αεροπορικές ε, εταιρείε. Δεν τα νοιάζει τα κατεμέλη γιατί δεν αφορά τον εθνικό προπολογισμό. Τα πληρώνουν οι επιβάτες των αεροπορικών γραμμών. Των αεροπορικών δηλαδή εταιρών, των αερομεταφορέων οι φορείς αυτοί ε, αντλούν τα εισοδήματά τους από μια μορφή ελέγχου της αγοράς μονοπωλιακή. Τα έχω μάθει τα μαθήματα αυτά. Η κυβέρνηση, αν ήταν υπόλογοι στο κοινοβούλιο, θα τους κυνηγούσαν οι βουλευτές που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά δεν είναι κυβερνητικό αυτό. Καταλαβαίνω κάποιες κυβερνήσεις να λένε ότι κάπως τα πράγματα λειτουργούν. Ούτε πέφτουν αεροπλάνα, ούτε προβλήματα έχουμε με τι εποπτικέ αρχέ, Οι συνδικαλιστικέ οργανώσει λίγο πολύ είναι ικανοποιημένε. α τα αφήσουμε όσο έχουν. Τι μα νοιάζει. Όχι, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται από τη σχετική νομοθεσία να επιτελέσουν σαφή πρόοδο για την ασφάλεια, τι δυνατότητες, την αποτελεσματικότητα προ το κόστο και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Κανεί δεν μπορεί να λέει ότι δεν θέλω να με κυνηγάνε οι συνδικαλιστέ. Όχι, αυτό δεν επιχείρημα. Βεβαίω και υπάρχουν ε, δυσκολίε που ε, δύσκολα ξεπερνούνται. Ένα παράδειγμα. Έχουμε να κάνουμε και με ένα πόλεμο, αν θέλετε, ιδεολογικό και οικονομικό. Οι Γάλλοι θέλουν δημόσια διοργάνωση των εποπτικών αρχών, Είναι οι Γερμανοί από ιδιωτικό φορέα. Ενώ στη Γερμανία συμβαίνει το αντίστροφο. ιδιωτική διοργάνωση με 100% δημόσια ιδιοκτησία. Κάποιοι χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα για να λένε δεν μπορούμε να συγχωνευτούμε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Και εγώ λέω όχι, λάθο. Διατηρήστε τι ιδεολογικέ σα διαφορέ, Αλλά παρόλα αυτά συναντηθείτε, συνεργαστείτε και σκεφτείτε τι δουλειά μπορούμε να κάνουμε από κοινού στο ΦΑΠ, Πώ μπορούμε να ενοποιήσουμε του πόρου μα. Ένα, ελεγκτέ ενέργεια κυκλοφορία, εκπαίδευση κοινή για όλου. Άλλοι που αναλαμβάνουν ε, την πληροφορική για όλε τι χώρε ανθρώπινοι πόροι για τι έξι χώρε. Μπορεί κανεί να γίνει πιο αποτελεσματικό λοιπόν και να συγχωνεύσει προσωπικό από διαφορετικέ ε, υπηρεσίε, από διαφορετικού φορεί και εταιρείε. Συνεργασία απαιτείται, αλλά απαιτεί αυτό και τα κρατημέλη και οι αερομεταφορεί να κάνουν αυτό το επιπλέον βήμα. Εκεί υπάρχει μεγάλη αντίσταση. Εκεί πρέπει να ενθαρρύνουμε του υπουργού. Μόνον οι υπουργοί μπορούν να δώσουν εντολέ. Δεν το δέχομαι να λέει ένα υπουργό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όχι. Είναι μέρος των ε, Υπουργείων οι εποπτικές αρχές. Όλες ε, εταιρείε παροχής υπηρεσιών είναι μέρος ε, του κράτους ή της δημόσιας διοίκησης ή 100% ελεγχόμενες από το κράτος. Δεν μπορώ να το δεχτώ λοιπόν. Τι μου λένε οι υπουργοί, δεν μπορώ να κάνω βήμα. Όχι, είναι θέμα πολιτικής τόλμης και πυγμής. Εάν δεν έχουν την πυγμή, Όπω σωστά είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή θα του προσάγει. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην κάνουν τη δουλειά του. Καμία. Ο Επίτροπος, εξ γνωρίζω, είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει. Αλλά τα κάτι μέλη αποφασίζουν. Και άλλε σύντομε απαντήσει γιατί περνάει ο χρόνο για τα προγράμματα επιδόσεων. Δύσκολο να πιεστούν τα κάτι μέλη εδώ, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί μόνο δει να ζητήσει αναθεώρηση. Εάν δεν γίνει κάτι, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Όμω υπάρχει μια έμεση δυνατότητα, δηλαδή λόγω τη νομοθεσία των ΦΑΜ εντό κάποιου FAB πρέπει να υπάρχει βέλτιστη χρήση των πόρων. Μπορεί να αναρωτηθεί λοιπόν κανεί τι εννοεί αυτή η έκφραση τι κάνετε με την βέλτιστη χρήση λόγου χάρη του συστήματός σας όσο χαζό κι αν είναι. Εδώ λοιπόν εναλλακτικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να προβλεφθούν. Και καλό είναι που τα παρακολουθεί στενά αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά να είμαστε επιφυλακτικοί. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να ετοιμάσει ένα νομοθετικό πακέτο SES e θα έπαιρνε τουλάχιστον ε, ένα χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο χρόνια με τη διαδικασία τη συναπόφαση, άλλο ένα χρόνο για τη μεταφορά, πενταετία συνολικά. Τέσσερα με πέντε χρόνια, δεν έχουμε τόσο χρόνο. Οι εκτελεστικέ αποφάσει τη Επιτροπή ε, για να ασκηθεί πίεση στα κάτι μελη είναι μια ιδέα. Αλλά εγώ είμαι ένα απαράδεκτο συνταγματολόγο ε, λόγω τη προηγούμενη σταδιοδρομία μου και ξέρω ότι τα πράγματα εδώ είναι πολύ δύσκολα. Λόγω χάρη, γερμανική γερμανικό σύνταγμα, εξαίρετο σύνταγμα, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο εδάφιο που λέει ότι η διαχείριση τη αεροπλοεία στη Γερμανία πρέπει να ε, από Γερμανού κυβερνητικού, κρατικού μάλλον φορεί ή προσθέθηκε πριν από δύο χρόνια με ευρωπαϊκά μέτρα, μέσω ευρωπαϊκών μέτρων. Τι θα πει ευρωπαϊκά μέτρα. Δεν είναι απόφαση τη Επιτροπή να αλλάξουν γερμανικοί κανόνε. Θα πρέπει να είναι απόφαση νομοθετών. Να είμαστε λοιπόν εδώ άκρος προσεκτική. Εάν σκεφτούμε τι θα λέγαμε στη γαλλική δίκηση με απόφαση της Επιτροπής. Δώστε μας όλες τις πληροφορίες που έχετε για, τα, για τη διαχείριση των ε, αερογραμμών. Ή σε μια ιδιωτική εταιρεία δώστε τα. Τι λέτε, θα τους άρεσε των Γάλλων. Τι θα λέγανε, οι εθνικέ μα πληροφορίε, η εθνική μα γλώσσα είναι κάτι που το μοιραζόμαστε με τον καθένα. Όχι, είναι δική μας, ε, δικό μα κυρίαρχο δικαίωμα. Ε, να το υπερασπιστούμε. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή πρέπει να είναι εδώ προετοιμασμένη και θα πρέπει να βγάλει τη μεράβδο τη μεγάλη και να ξέρει πότε θα τη χρησιμοποιήσει. Διότι αν υπάρξει προσαγωγή στο ΔΕΚ, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Θα μπορεί να επιβάλλονται ημερήσια πρόστιμα. Κάποιοι Γερμανοί υπουργοί φαίνεται να μην το σκέφτηκαν, αλλά τώρα βλέπουν τι καραδοκεί. Λοιπόν, δεν θέλουμε σύγκρουση εδώ. Δεν θέλουμε κατά μέτωπο σύγκρουση. Καλέ σχέσει επιδιώκουμε. Γι' αυτό δεν απειλούμε τα κράτη-μέλη. Κίνητρα θέλουμε να του δώσουμε. Τα ενθαρρύνουμε. Γι' αυτό και ο αντιπρόεδρο Κάλλα νομίζω θα πρέπει να στείλει προειδοποιητικέ επιστολέ. Δεν θα τι έλεγα προ-διαδικασίες παραβάσει επιστολέ που προηγούνται δηλαδή αυτή τη διαδικασία. Όχι, προειδοποιητικέ είναι. Και από τα καλά παραδείγματα να διδαχθούμε ότι υπάρχει δυνατότητα δημιουργία αποτελεσματική στο Φαμπ και δεν αποτελεί, δεν υπάρχει λόγο να μην δημιουργηθούν τα υπόλοιπα FAB όπω πρέπει, να μην διοργανωθούν όπω πρέπει. Και να ολοκληρώσω, γιατί βλέπω ότι ο πρόεδρο κοιτάει το ρολόι του, για τη Βόρεια Ιταλία δεν ξέρω, θα πρέπει να ενημερωθώ. Για το FAB CE Κεντρικής Ευρώπης θα είμαι την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, θα δω τι γίνεται με αυτό το FAB της Κεντρικής Ευρώπης. Ε, δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να πω τίποτε ακόμη. Το δυσκολότερο νομίζω ότι θα είναι αυτό της γαλάζιας Μεσογείου, το Med. Για διάφορους λόγους, έτσι, το πιο δύσκολο να μένετε να είναι. Ελπίζω ότι θα έχουμε λειτουργικά τμήματα ενέργειο χώρου που να λειτουργήσουν τελικά. Θα τα έχουμε. Μη λέτε δεν θα γίνει. Εγώ νομίζω ήδη λειτουργεί σε έναν βαθμό. Οι Βρετανοί και οι Ιρλανδοί και οι Δανείοι Σουηδοί πάρα πολύ καλά τα πάνε ήδη. Ναι, η δικιά σα ομάδα, η ομάδα του Δούναβη, μπορεί να λειτουργήσει ω το Δεκέμβρη. Άντε. Και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε καλό δρόμο. Νομίζω λοιπόν ότι με λίγη με λίγο σπρόξιμο και το ΦΑΜΠΕΚ μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο. Τώρα, γιατί δεν προχωράει η κεντρική Ευρώπη, γιατί υπάρχει και τέλμα, θα το ανακαλύψω, για να είμαι ειλικρινής. Και τα υπόλοιπα τέσσερα Φάμπεκ, όμως, εφικτά είναι. Και αυτό τη βαλτική Πολωνία, Λιθουανία. Δεν βλέπω λόγο δύο μικρέ. Τέλο, πάντων, μια μεγάλη και μια μικρή, για να μην προσβαλώ και κανέναν. Να μην μπορούν να συνάψουν μια κρατική συμφωνία. Ελπίζω επίση και αυτό το νοτιοδυτικό θα λειτουργήσει. Βλέπω λοιπόν να υπάρχουν θετικέ προοπτικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προχωρήσει το όλο θέμα. Είναι σημαντικό για την ομάδα Α6. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο. Δεν το έχω και σίγουρο διότι μιλάμε για μέσοπρόθεσμες ή και μακροπρόθεσμες εξέλιξεις. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορούν να πάνε και να μας διευκολύνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει να κάνει το Κοινοβούλιο, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να στηρίξει, να ενθαρρύνει την Επιτροπή ώστε να στηρίξει με τη σειρά της τα κράτη-μέλη. Και σας παρακαλώ, όπως είπε και Ζήνε, πηγαίνετε στο κοινό, μιλήστε στις αερογραμμές και στους υπευθύνου τους. Φροντίστε και το κοινό να ενδιαφερθεί για το θέμα. Χρειαζόμαστε πίεση, να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη, όχι μόνο από την Επιτροπή και από τι αερογραμμέ και από τον βιομηχανικό κλάδο. Δεν το κάνουμε αυτό μόνο και μόνο για λόγου νομικήστικου. Για τον επαγγελματικό κλάδο το κάνουμε, για του πολίτε. Η ευαισθησία λοιπόν, η ευαισθητοποίηση του κοινού για όλο το όλο θέμα θα είναι σημαντική. Και αν κάτι ξέχασα, να μου στείλετε email. Θα τα απαντήσω. Ευχαριστώ. Well, thank you very much, George. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Πάντοτε με χαρά ε, σε βλέπουμε και περιμένουμε και την έκθεσή σου την επόμενη, ξέροντας ότι θα είσαι λίγα δραστήριος μέχρι το Δεκέμβριο, θα καταβάλεις κάθε προσπάθεια να προωθήσεις το θέμα. Ό,τι μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε θα το κάνουμε και η Κομισιόν επίσης. Θα χαρούμε να σε ξαναδούμε την, και να μάθουμε τα νεότερα την επόμενη φορά και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. we just got to rearrange the table now. Πρέπει τώρα να αναδιατάξουμε το Προεδρείο εδώ. Okay, colleagues, if Λοιπόν, συνάδελφοι, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε με το επόμενο θέμα, που είναι η κοινή συνεδρίαση με τη δική μας Επιτροπή και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Παρακαλώ να ηρεμήσει το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Μάλκομ Χάρμπερ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς που είναι μαζί μας σήμερα. Έχουμε μια ξεχωριστή μερίσια διάταξη γιατί είναι κοινή συνεδρίαση. Είναι καταρχάς ανακοινώσει του Πρόεδρου, μετά παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης, ε, ε, σχέδιο πρωτοβουλίας, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας επόμενη συνεδρίαση κλπ. Λοιπόν, συμφωνείτε με την μερίσια διάταξη της κοινή συνεδρίασης, ωραία, και μπορούμε να προχωρήσουμε με τον Μάλκομ. Η καινούρια η υπηρεσία του e-call καλύπτει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του IMCO και Τρανσκο και επίσης Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλή ιδέα να καλυφθούμε από την διαδικασία του άρθρου 51, του κανονισμού, του άρθρου 51 του κανονισμού. Και γι' αυτό ακριβώς ισχύει, θα ισχύσει το άρθρο 51 του κανονισμού στο σχέδιο γνωμοδότησης ιδίας πρωτοβουλίας. Οι συντονιστές έχουν συντάξει μία κοινή έκθεση την οποία θα εξετάσουμε και η οποία θα ψηφιστεί ε, και από τις δύο επιτροπές υπό την κοινή προεδρία. Ε, τα ε, δικαιώματα τα οποία ανήκουν στις αρμοδιότητες κάθε επιτροπής μπορούν να ασκηθούν μόνο όταν οι επιτροπές αυτές συνεδριάζουν από κοινού και αυτή τη στιγμή την Προεδρία και την αίθουσα την έχει η Τράνσκο, την επόμενη φορά μπορεί να είναι η ΙΜΚΟ. Ε, μπορεί να ε, μιλήσει, να μιλήσει όποιος ε, επιθυμεί και από τις δύο επιτροπές. πρέπει να το ξέρουν, αν δεν το ξέρουν μπορεί να μην μιλήσουν καθόλου. Λοιπόν, ε, απλώς ε, ορισμένες, ε, ορισμένα διαδικαστικά σημεία ήθελα να διευκρινίσω για να ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ. Ο κύριος Χάμπερ. Um, Ευχαριστώ. Είναι μια, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά, διότι προερχόμενοι από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες αναγνωρίσαμε την ανάγκη μιας κοινή προσέγγισης σε αυτήν τη γνωμοδότηση, ιδίως σε θέματα ε, στρατηγικής, πολιτικής και νομοθεσίας. Από πλευράς τώρα ε, Επιτροπής Μεταφορών, ε, η αρχή είχε γίνει με την οδηγία για τις ενιαίες υπηρεσίες και την ηλεκτρονική επικοινωνία όπου είχαμε επισημάνει ορισμένη την ανάγκη να υπάρξει ένα αριθμό κλήση ε, για τις, την προσφορά αυτών των ε, ενιαίων υπηρεσιών, το 112. Εν συνεχεία είχαμε συντάξει μια έκθεση για την ε, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα και δυνατότητα κλήσης αυτού του αριθμού και δεδομένου ότι συζητούμε πάντοτε ηλεκτρονικά δίκτυα, το θέμα αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή Μεταφορών. Τώρα από το δικό μου υπόβαθρο, ο, όταν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής ο Επίτροπος Λίκανεν το 2003 είχαμε ασχοληθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητιστών και είχαμε τότε συγκαλέσει ένα φόρουμ, μια ε, συνεδρίαση για το ε112 και είχε ακουστεί τότε για πρώτη φορά η πρόταση. Υπάρχει λοιπόν εδώ και χρόνια. Η πρόταση λοιπόν αυτού του e-call, ε, της ε, κλήσης, δεν είναι μια καινούργια πρόταση, αλλά ε, έχει συζητηθεί επί μακρόν και είναι ένα ωφέλιμο μέτρο που θα σώσει ζωές ε, και θα προλάβει ατυχήματα και θανάτους ε, στις χώρες μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για τη συνεργασία και ελπίζω μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Θέλω να αρχίσω με τους δύο συγητές, πέντε λεπτά ο καθένας. και συνεχεία θα ζητήσω την εισηγήτρια από, από πλευράς ΙΜΚΟ να μιλήσει πρώτη και συνεχεία ο συνεισηγητής από πλευράς Τράνσκο και εν συνεχεία η σκιώδης εισηγητής και έτσι ακριβώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς και εκ μέρους ε, της ΙΜΚΟ η Όλγα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στις αρχές της χρονιάς είχαμε μία ακρόαση για το θέμα αυτό, για αυτήν την προβληματική. Τροποποίησαμε τις διαδικασίες και χαίρομαι που σήμερα μπορούμε και βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια το σχέδιο έκθεσης το οποίο θα σας υποβάλουμε από κοινού με τον συνάδελφο Κόχ. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι συμφωνούμε για την αρχική ιδέα της έκθεσης αυτής. Το σύστημα αυτό, e-call, πρέπει να γίνει ένα γενικευμένο σύστημα και θα πρέπει να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί το νούμερο αυτό 112 και να βασίζεται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και να μπορεί κανείς από όλα τα οχήματα, από οπουδήποτε, να μπορεί όσο γίνεται καλύτερα τόσο για τους οδηγούς όσο και για όλους όσους βρίσκονται σε κυκλοφορία. Πρέπει να είναι δωρεάν το νούμερο αυτό και να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες. Μια από τις κύριες προϋποθέσεις είναι τα κέντρα ΠΕΣ και ΑΠΕ. Εδώ είναι τα κράτη-μέλη τα οποία πρέπει να φροντίσουν τα κέντρα αυτά να μπορούν να διαχειρίζονται όλες τις επίγουσες αυτές κλήσεις. Πρέπει να δούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος σε κάθε χώρα. Σήμερα στην αγορά υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που δεν λειτουργούν όμως όλες τις χώρες και προτείνονται μόνο για τα πολυτελή οχήματα. Το μερίδιό του στην αγορά είναι πολύ αδύναμο ακόμα. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Το e-call λοιπόν πρέπει να μπορεί να λειτουργεί μέσα στο 112. Το σύστημα e-call αρχίζει να λειτουργεί από τη στιγμή που γίνεται μια έκτακτη κλίση και ο καταναλωτής πρέπει να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει προστασία των προσωπικών ε, δεδομένων και στην περίπτωση του e-call αλλά και στην περίπτωση άλλων ιδιωτικών αντίστοιχων υπηρεσιών. Η διαλειτουργική πλατφόρμα θα οδηγήσει κατά τη γνώμη μας στη στήριξη της καινοτομίας και στην αύξηση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, του ευρωπαϊκού κλάδου. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο έτσι ώστε μέχρι το 2015 να έχουμε αυτό το σύστημα, να μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε το e-call μέσα από το νούμερο 112. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Από το 2002 έχουμε αρχίσει να το σκεφτόμαστε αυτό. Και το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει κάποιες προτάσεις ρύθμισης εφόσον η σεθελοντική βάση πρόσβαση δεν λειτουργήσει. Το 2011 η κυρία Κρέσ παρουσίασε ε, κάτι σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας ζήτησε να φροντίσουμε να υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα αυτό e-call της ηλεκτρονικής κλίση δηλαδή, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί έτσι σώζονται ζωές. Και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέλει αυτό. Δυστυχώς πέρσι όμως δεν επιτέχθη καμία πρόοδος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό και εγώ σήμερα απευθύνομαι στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ρωτάω ποια είναι η γνώμη τους σήμερα. Γιατί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει κανένα σχέδιο για τα ε, τυποποιημένα ε, οχήματα στην Ευρώπη, ενώ έπρεπε να το έχει κάνει κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της χρονιάς αυτής. Πότε θα ξεμπλοκαριστεί η κατάσταση και πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φέρει σε πέρας ε, τις υποχρώσεις, τις υποχρώσεις που έχει ήδη ε, αναλάβει νωρίτερα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα. Όσον αφορά τις τροπολογίες, 8 Μαΐου προτείνουμε να είναι η προθεσμία με τον συνάδελφο Κοχ. Θα συνδρεθούμε και θα εξετάσουμε τότε όλες τις τροπολογίες και θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 19 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τώρα φαντάζομαι ότι ο συνάδελφος Κόχ θα πάρει το λόγο. Του δίνω τη σκητάλη και περιμένω τις τροπολογίες σας και από τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ. Η πρόταση αυτή μου φαίνεται ότι έχει μακρά ιστορία. Πριν από 10 χρόνια μίλησα και εγώ πρώτη φορά στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Σεναλόβα για την, ε, τη σαφή της, ε, τη σαφή της παρουσίαση και ευχαριστώ και τους τειώδη εισηγητές που συνδέονται με αυτό το θέμα επίσης ε, από καιρό. Έχουμε κοινέ απόψεις σε ένα σημαντικό θέμα και κοινού στόχου, Ο στόχος είναι ένα λειτουργικό e-call που θα σώζει ανθρώπινες ζωές, ένας αριθμός που θα είναι προσβάσιμος σε όλους, που θα λειτουργεί σε όλα τα σημεία παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα e-call που θα διευκολύνει και την ιατρική βοήθεια με στοιχεία δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών. Αυτό, αυτή η υπηρεσία θα είναι σημαντική και στους χώρους εργασίας και στις επιχειρήσεις και στις ασφαλιστικές εταιρείες και στις ε, αρχές αστυνομικές και άλλες. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μία ενιαία υπηρεσία η οποία θα προσφέρεται δωρεάν σε όλους. Και επί εθελοντικής βάσεως μπορούν ή e-call ανάλογα με το τι προσφέρει ο δημιουργός να συμπληρώνουν το δίκτυο. Ε, το η επιτυχημένη λειτουργία του e-call αυτού το 112 ε, εξαρτάται από την καλή επιλογή του λογισμικού. Εάν αυτό αποδειχθεί σωστό όλα τα άλλα θα λειτουργήσουν καλά όπως τα θέλουμε. Τώρα θα πω λίγα λόγια για το πώς θα λειτουργήσει το όλο ε, για να παρακινήσουμε και τον ε, ευρωπαϊκό οικονομικό και βιομηχανικό τομέα να ε, δείξει μια ε, διεθνή πρωτοβουλία και να πρωτοπορία. Καταρχάς θα χρειαστεί μια, ένα, μια έκθεση η οποία ήδη έχει αποφασιστεί να συνταχθεί Αλλά από ποιον θα γίνει αυτή η έκθεση. Υπάρχει ένα καινούργιο χρονοδιάγραμμα για, μία, για έναν τέτοιον κανονισμό που θα καλύπτει αυτό το equal. διότι η οδηγία για τις έξυπνες μεθόδους μεταφορών ήδη υπάρχει. Πρέπει τώρα να βρούμε και τον κανονισμό στον οποίο θα εμπίπτει αυτό το δίκτυο. Επίσης πρέπει να βρούμε και ένα κατάλληλο κείμενο το οποίο θα καλύπτει και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και όχι μόνο τους ε, κατασκευαστές ασύρματων δικτύων και άλλων τεχνολογικών υπηρεσιών. Τρίτον, η κυρία Γκρές, η κυρία Επίτροπος, είπε τον παρουσίασε το e τον ε, προηγούμενο Σεπτέμβριο και έδειξε έτσι ιδιαίτερο ενθουσιασμό να υποστηρίξει την πρόταση αυτή όπως και εμείς. Τώρα ο Επίτροπος Ταγιάννης στις 8 Μαρτίου μας παρουσιάζει ένα μορατόριο και λέει θα σταματήσουμε όλες τις ρυθμίσεις, ε, όλες ε, τις, ε, όλα, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα προς όφελος των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Πρέπει να πω ότι, ότι ε, τρόμαξα με αυτά τα οποία άκουσα, ε, διότι εδώ προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάτι τα οποία θα, θα, θα, θα σώσει ανθρώπινες ζωές ε, ή θα προλάβει τέλο πάντων ατυχήματα και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μορατόριο το οποίο, δεν, το οποίο δημιουργεί εμπόδια στην παροχή αυτών των υπηρεσιών και θα βλάψει αυτό το μορατόριο όλους τους πολίτες μας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε ότι το δίκτυο αυτό, οι κλήσεις αυτές, το 112, θα είναι προσβατό σε όλους, θα είναι δηλαδή δημόσια τα δεδομένα και προσβάσιμα σε δημόσιες αρχές. Και ε, σε μία από τις προηγούμενες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα ζητήσει η Κομισιόν να σκεφτεί επίσης ε, παρόμοιους αριθμούς ε, άμεσης κλήσης για φορτηγά και για μοτοσυκλέτες. Τώρα το θέμα της ρύθμισης των προσωπικών δεδομένων μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και μπορούμε ε, να βελτιώσουμε και την ε, παραγωγή των, ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας εάν συμφωνήσουμε στον κοινό σκοπό. Ισκιώδης. Τώρα την κυρία Χολουστάν δεν τη βλέπω. Η κυρία Γκουρμάη τότε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που βλέπω δύο τόσο εξαίρετους προέδρους τον έναν δίπλα στον άλλον. Ήταν πολύ καλός φίλος ο άλλος πρόεδρος σε μένα, με έχει βοηθήσει στην πρώτη μου έκθεση πάρα πολύ. Είναι καλό που συνεργάζονται οι δύο επιτροπές μας. Έχουμε και συμπρόεδρους και συνεισηγητές. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που μπορούμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό σήμερα. Νομίζω ότι πριν καταλήξουμε σε μια ενιαία έκθεση, καλό είναι να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Συμφωνώ όμως είπαν οι συνάδελφοι. Εννοείται, ε, αφού μπορούν να σωθούν οι ζωές, πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Ε, όταν ε, είχαμε σαν αριθμό ότι 40.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους, ξέραμε ότι 4.000 θα είχαν σωθεί αν υπήρχε αυτό το σύστημα. Φυσικά και πρέπει να τα δώσουμε τα χρήματα που χρειάζεται γι' αυτό, γιατί η κρίση υπάρχει, οι κρίσει έρχονται και παρέρχονται, οι ανθρώπινε ζωέ όμω πρέπει να σώζονται. Το πρόγραμμα δράση για την, ασ... την οδική ασφάλεια ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Κοφού ήταν ο σκιώδης μου τότε. Και με αυτόν τον τρόπο όμως θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο διαλειτουργικό e-call μέσω οδηγίας. Πρέπει να είναι δικαίωμα του καταναλωτή και προστασία του καταναλωτή η πρόσβασή του από παντού γεωγραφικά στο e-covel. Άρα η γεωγραφική κάλυψη πρέπει να είναι πλήρης. Χαίρομαι λοιπόν για την συνάντηση αυτή. Απ' την άλλη μεριά όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων πρέπει να κατανοήσουν ότι όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους πρέπει να έχουν την τεχνική υποδομή να αναγνωρίζουν το σήμα του e και να έχουν και τον εξοπλισμό που χρειάζεται το κάθε όχημα για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στο e-call και να μην πρέπει κανείς να το πληρώσει έξτρα αυτό. Επίσης το e πρέπει να είναι και εύχριστο αλλά και κόστος που να μπορεί να επομιστεί ο καταναλωτής που αγοράζει το αυτοκίνητο. Τώρα, η εθελοντική βάση δεν πιστεύουμε ότι φτάνει. Ήταν ανεπαρκής. Υπάρχει από το 2003 και ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση προκειμένου και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία να υπογράψουν το ε, memorandum, το μνημόνιο. Ξέρω βέβαια ότι δεν είναι αυτή η πρώτη ανησυχία του Σερκοζή σήμερα, Πάντως, αν δούμε τι έχουμε ήδη, έχουμε την νομοθετική δράση που προέβλεπε τρία μέτρα, Έχουμε τη σύσταση της Επιτροπής που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο που ζητά από τα κράτη-μέλη να διασφηνίσουν ότι οι υπάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα φροντίσουν να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στο e-call. Έπειτα Μέχρι τα τέλη της χρονιάς πρέπει να υιοθετηθούν οι κατεξοδότηση πράξεις, είναι στο χέρι μας δηλαδή, και υπάρχει και η πρόταση νομοθετική στο τραπέζι. Άρα έχουμε όλες τις ιδέες για την βελτίωση. Ας ε, ξεκαθαρίσουμε, όταν δύο δυνατές επιτροπές συνεργάζονται, τίποτα δεν μπορεί να είναι αδύνατον. Ευχαριστούμε κυρία Παβάνοβα από την ΙΜΚΟ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ του δύο πρόεδρους μας που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Έτσι μπορούμε να διοργήσουμε μια καλή μέθοδο συνεργασία. Και για πολλά άλλα θέματα θα μπορούσαμε να εξακολουθήσουμε αυτή την τακτική. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για το έργο τους επί των θεμάτων αυτών. Συνολική και διεξοδική η γνωμοδότηση και τοποθέτηση για τι νέε υπηρεσίε που θα προβλεφθούν μέσω του e-call, όμως κάποιες ιδέες που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση και καλό θα ήταν, καλό θα ήταν να του δοθεί έμφαση. Εδώ μιλάμε σήμερα για ένα σύστημα που λίγο πολύ συγκριτικά με το πόσο γρήγορα προχωρούν τα λογισμικά, οι τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά, τουλάχιστον μιας δεκαετίας ηλικία. Δηλαδή, Μα προσχολεί και η αποτελεσματικότητα ω προ το κόστο, αλλά και η αποδοτικότητα. Επίση, η ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Για την εγκατάσταση και την χρήση του συστήματος. Τι καλούς λόγους να βρούμε. Δεν υπάρχουν λογικές εξηγήσεις για το πόσα οδικά ατυχήματα έγιναν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς υποδομέ ή κάλυψη κινητής τηλεφωνίας ή τέλο πάντων από παροχή κινητή τηλεφωνίας. Πόσα από αυτά θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί στην πράξη. Θα μπορούσε κανείς να τηλεφωνήσει στα επίγοντα εγκαίρως σε αυτές τις αποκλεισμένες περιοχές και πώς από αυτά θα προλαμβάνονταν επειδή ούτως ή άλλως μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Η καθυστέρηση της κλίσης ήταν σημαντικός παράγοντας επιδείνωσης της κατάστασης. Δεν τα έχω δει αυτά και τα βρίσκω ζωτική σημασία. Επίση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι υποδομέ των κατώμελών έχουν ε, δημιουργηθεί. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει για τα e-call και επίσης το σύστημα 112. Σε καποια κρατημέλη υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για ιατρικές κλήσεις λόγου χάρη. Μία στις τέσσερις φαίνεται να αποδίδει. Εάν πέραν αυτών των προβλημάτων τα συσχετίσουμε και με ένα άλλο σύστημα, μπορεί τελικά να τα επιτείνουμε τα προβλήματα αντί να τα επιλύουμε. Επίσης, η τεχνολογική ουδετερότητα είναι ένα ζήτημα καθοριστικής σημασίας. Για την αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και την αποδοτικότητα του συστήματος χρειαζόμαστε νέες ευκαιρίες για τις εταιρείε. Να μπορέσουν να αναπτύξουν δηλαδή πιο σύγχρονα μέσα που να είναι συμβατά μεταξύ τους και να δώσουμε και στον κλάδο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα δυνατά μέσα, τεχνολογικά μέσα. Να επαναλάβω ότι εγώ στηρίζω την πρόβλεψη ενό πανευρωπαϊκού συστήματο e αλλά προηγουμένω να βεβαιωθούμε ότι όλε οι σημαντικέ μα μέρημνε έχουν καλυφθεί. Ιδίω ό,τι αφορά τι υποδομέ. Και προτού ζητήσουμε την υποχρεωτική εφαρμογή για όλε τι περιπτώσει ηλεκτρονικών κλήσεων. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μπένιον για την Επιτροπή Μεταφορών. Έχουν ε, φυγεί κάτι από τα θέματα που ήθελα να καλύψω. Και σε πρώτη φάση να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την πολύ καλή τους έκθεση που καλύπτει ζητήματα όπως η προστασία των δεδομένων, η στάυρωση με ιδιωτικέ υπηρεσίες. Όμως εδώ θέλω να κάνω και εγώ τις παρατηρήσεις. Το βασικό ζήτημα παραμένει. Υπάρχει διχογνωμία εδώ μεταξύ της ανάλυσης αποτελεσματικότητας του κόστους και της αναλογίας αποτελεσματικότητας του κόστου. κόστους. Δαπανούμε σωστά τα χρήματά μας, ε, τα κονδύλια που προβλέπονται ή μπορούμε να βελτιώσουμε με άλλους τρόπους την οδική ασφάλεια, έστω και με το ίδιο κόστος. Θα ήθελα λοιπόν εδώ μία πιστική ανάλυση κόστους ωφελίας. Προτού δεσμευτούμε. Προτού δεσμευτούμε για το εγχείρημα αυτό. Επίσης, ε, έγινε συζήτηση για το κατά πόσον οι νομαδικές συσκευές μεγάλων αποστάσεων θα μπορούσαν να καλύπτονται. Εάν επιτρέψουμε ένα τέτοιο σύστημα και αυτές οι συσκευές δεν χρησιμοποιηθούν, σε 8-10 χρόνια δεν θα έχουν εξοπλιστεί ακόμη όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε η αποδοτικότητα προς το κόστος, η σχετική δηλαδή αναλογία θα είναι πολύ χαμηλή. Πρέπει να τους επιτρέψουμε τις συσκευέ αυτές, ε, διότι το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ ψηλό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εδώ μόνο τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί μετά την ημερομηνία υλοποίηση. Επίσης, συμφωνώ ότι η Επιτροπή μας πρέπει να είναι τεχνολογικώς ουδέτερη. Εάν προχωρήσουμε με το σύστημα αυτό, θα πρέπει να είμαστε ελαστικοί. Όλες οι τεχνικές βελτιώσεις να μπορούν να καλυφθούν εφόσον χρειάζεται. η αλυσίδα διάσωσης και το κατά πόσον θα πρέπει να έχει ε, εγκατασταθεί προτού την εκκίνηση του συστήματος. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε μέχρι το 2015, είναι εφικτό και είναι και πολύ σημαντικό. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ανεπαρκής απόκριση. Αυτό έχει να κάνει και με την αναλογία κόστους ωφελίας που ανέφερα προηγουμένως. Εδώ θα πρέπει να βεβαιωθούμε τι κάνουμε. Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση και δουλειά. Ο αριθμός ανεπαρκών αποκρίσεων δεν επιβάλλει τη χρήση των επιγόντων επικουσών υπηρεσιών μάλλον. Δεν φαίνεται ότι θα είναι η δαπάνη ανάλογη με το κόστος που εμείς προβλέπουμε. Πόσο χρόνο θα χρειάζεται για να κινητοποιηθούν τα επίγοντα για ίσονο σημασία περιστατικά που τώρα δεν καλύπτονται και πόσο χρόνο θα χάνεται εφόσον οι ηλεκτρονικέ κλήσει πρέπει να κατευθυνθούν αλλού και τα ασθενοφόρα τελικά είναι απασχολημένα με τα ίσονο σημασία ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν η φωνητική επαφή να γίνεται ταχύτερα και να είναι και αποτελεσματική ώστε να αποφεύγονται οι ανεπαρκείς αποκρίσεις, δηλαδή οι άστοχες αποκρίσεις. Ευχαριστούμε ο κύριο Τέιλορ για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι το σύστημα θα μπορούσε να είναι μια θετική συμβολή, συμβολή προς την ασφάλεια. Αλλά με άλλα μέτρα μαζί που θα έπρεπε να επιβληθούν, ώστε να περιοριστεί η ταχύτητα και η κατανάλωση αλκοολούχων αυτοί είναι οι δύο βασικότεροι κίνδυνοι για το επιβατικό κοινό και τους κατοίκους επίση. Όσους δεν επιβαίνουν σε οχήματα δηλαδή. Μια τεχνική τώρα παρατήρηση για τις επίγουσες υπηρεσίες. Θα πρέπει να αποστέλλονται οι σωστές πληροφορίες με τη σωστή σειρά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα φωνητικής επαφής με τους ε, επιβάτες του οχήματος ή με τους οδηγούς. Αυτό θα ήταν πραγματικά χρήσιμο. Πρέπει κάτι τέτοιο να ισχύσει. Όσοι λοιπόν αναπτύξουν αυτά τα συστήματα θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι λειτουργούν αποτελεσματικά και να εξοπλίσουν σωστά τα οχήματα. Το κοινό PSAP είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να το αναθέσουμε εξ ολοκλήρου σε ιδιώτε Το λέει όμω και η έκθεση στο τμήμα για την προστασία των δεδομένων. Εκεί χρειάζεται κάποια προσαρμογή. Μεγαλύτερο βαθμό προστασία θα χρειαστούμε κατά την άποψή μα. Τέλο, το ζήτημα παραμένει για το κόστος. Οι υποδομές πόσο θα κοστίσουν. Ποιο θα καλύψει το κόστος αυτό. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το μελετήσουμε διεξοδικά και μετά να συμφωνήσουμε κιόλα. Διότι ένα είναι να λέμε ότι θα δημιουργήσουμε το σύστημα και άλλο να εξηγήσουμε πώς θα χρηματοδοτηθεί. Η παραγωγή. βεβαίως θα κοιτάξουν να πετάξουν το μπαλάκι του κόστους ε, στην τιμή του οχήματο στον καταναλωτή. Αυτό λογικό είναι. Εάν σκεφτείτε πώς θα ήταν ένα όχημα χωρίς ζώνες ασφαλείας, θα καταλάβετε γιατί στο μέλλον κάποτε θα είναι δύσκολο να πουληθεί και ένα όχημα χωρίς e-call, ηλεκτρονική κλίση. Θέλουμε λοιπόν εφη οχήματα μένα, αλλά σημαντικότερο είναι να έχουμε και ευφύς οδηγούς. Όσο πιο σύντομα λοιπόν να απτύξουμε την ευθεία των οδηγών, τόσο καλύτερα. Ευχαριστούμε. Η ευθεία των οδηγών είναι το βασικό πρόβλημα, ούτως ή άλλως. Η κυρία Ντρόσπακ, για τους ε, συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, ώστε να δούμε και το αυτοματοποιημένο όχημα του μέλλοντος. Πολλές ε, είναι οι φάσεις μέχρι να καταλήξουμε και, και αυτή είναι μια από αυτές. Τέλος πάντων, πέρα από τα αστεία, νομίζω είναι σημαντικό που έχουμε αυτήν την κοινή έκθεση από τις δύο επιτροπές. Το εκτιμώ ιδιαίτερος, εκτιμώ την ε, συνεργασία μας σε τέτοια ζητήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ξανά. Κάποιες εταιρείε ήδη συμπεριλαμβάνουν το σύστημα αυτό στα οχήματά τους. Η Peugeot, η Volkswagen. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τόσο δαπανηρό και περίεργο σύστημα. Ήδη στα Πασάτ χρησιμοποιείται. Όμως έχουμε ακόμη δρόμο να κάνουμε. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σύστημα, εάν θέλουμε να το προκρίνουμε. Και χρειάζεται και καλύτερη διασύνδεση, εάν θέλουμε να λειτουργεί αποτελεσματικά. Θα πρέπει να λειτουργεί δηλαδή ένα τέτοιο σύστημα παντού. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η επιβολή. Αλλά καταλήγουμε πάλι στο εξή σημείο. Πού ε, τελειώνει η προσωπική ελευθερία και πού αγγίζει την προστασία των δεδομένων. Τελικά μας παρακολουθεί ο μεγάλος αδερφός όταν οδηγούμε. Αυτό θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε. Ή μπορούμε να τον πετάξουμε από πάνω μας. Θα πρέπει λοιπόν να Μα απασχολήσουν και οι λεπτομέρειες. Ποιοι θα αποκρίνονται στις κλήσεις, η αστυνομία, ένα νοσοκομείο, ποιο απαντά εφόσον αποσταλεί μήνυμα. Εάν λοιπόν ανοίξουμε θέματα προς τη ζήτηση για το άμεσο μέλλον, θα πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Δεν θα επαναλάβω όλα τα θετικά σχόλια που ακούσαμε στους συναδέλφους, απλώς θα πρέπει να δείξουμε τη δέουσα προσοχή. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος Χάρμπορ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ως και όδης για την ομάδα, για, ναι, εκ μέρου τη ομάδα μου παίρνω το λόγο για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πρώτον, ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια και τον εισηγητή για τη δουλειά τους. Είναι ένα πρώτο βήμα και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να ξανανοίξουμε κάποια από τα ζητήματα που μας απασχολούν και που έχουμε στο μυαλό μας εδώ και πολύ καιρό. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι κάτι γενικότερο όσον αφορά τις οικουμενικές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες. Θέλω να σας επενθυμίσω από την οδηγία σας λέω τώρα, σας διαβάζω τώρα, για τις οικονομικές ε, οικουμενικές υπηρεσίες και είναι κάτι το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή μας το 2009. Λέει, τα κράτη-μέλη θα διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας θα ε, προσφέρουν πληροφορίες για τις κλήσεις ε, δωρεάν ε, σε περιπτώσεις εκτάκτων κλήσεων εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες. Αυτό ισχύει για το 112 και λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επεκτείνουν την υποχρέωση και σε άλλα εθνικά νούμερα έκτακτης κλήσης. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο για τα αυτοκίνητα το σύστημα. Αν εσείς από το κινητό σας πάρετε το 112 θα πρέπει η τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε να πηγαίνει ως ένδειξη στις υπηρεσίες του 112 που καλείτε. και αυτό πρέπει να γίνεται και από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, μερικές φορές τη δυνατότητα αυτή τη χρησιμοποιούν ε, οι υπηρεσίες ε, έκτακτης ανάγκης. Δεν το έχουν όμως όλοι. Και ελάχιστη πρόοδος έχει γίνει. Γι' αυτό και έρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Παρβάνοβα, δηλαδή το θέμα της τεχνολογίας. Γιατί τώρα είναι να συμφωνήσουμε για την τεχνολογία, δηλαδή την τοποθεσία και να μπορεί κανείς να έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει το κινητό του θέλει, αλλά να μπορεί να υπάρχει αυτή η ένδειξη τοποθεσίας. Για το χειρισμό των κλήσεων, το σύστημα e-call στο χήματα θα χρησιμοποιεί βασικά το ίδιο σύστημα το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει παντού στην περίπτωση που καλούμε το 112, αναγνώριση τοποθεσία δηλαδή. Τώρα το θέμα του ιδιωτικού βίου πρέπει να μπορεί κάποιο και γίνεται αυτό. Να μην υπάρχει αυτή η ένδειξη. Αν δηλαδή κάποιο δεν θέλει όταν α, ε, τηλεφωνήσει στο 112 να φανεί το που βρίσκεται, μπορεί να το κάνει. Να βγάλει αυτή την εφαρμογή δηλαδή. Πάντως θέλω ευχαριστήσω την κυρία Βάνοβα η οποία φρόντισε και ήρθε σε επαφές ε, από την Πράγα με αρμόδιους για τα θέματα δικής ασφάλειας που ήρθαν και μας μίλησαν. Υπάρχουν κάποιες διαφάνειες επίσης που μας ε, έδωσαν και ίσως οι συνάδελφοι θα πρέπει να τις κοιτάξουν. Τώρα, τα οχήματα. Το θέμα της τοποθεσίας ε, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τα οχήματα και θα είναι πιο εύκολο όταν είναι σε ανοιχτό χώρο. Το άλλο τώρα είναι ε, το θέμα των αερόσακων. Μήπως όταν ανοίγει ένα αερόσακο, τότε μπορεί να πηγαίνει το σήμα για την τοποθεσία. Ο αρμόδιο από την Πράγα είπε ότι χρησιμοποιούν αυτήν την πληροφορία για να αντιληφθούν πόσο σοβαρό είναι το ατύχημα και είχε να μας πει και άλλα για την κατεύθυνση που παίρνει το όχημα, αν έχει βγει από τον αυτοκινητόδρομο, αν είναι πολλαπλό το ατύχημα, βλέκονται δηλαδή πολλά οχήματα, πόσο σοβαρό είναι το ατύχημα για να κρίνουν πώς πρέπει να αντιδράσουν. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που είναι διαθέσιμοι σήμερα θα βοηθήσουν πάρα πολύ τις υπηρεσίες έκτακτες ανάγκες και θα τις κάνουν να αντιδράσουν πιο αποτελεσματικά. Βέβαια τίθεται το θέμα του κόστους και η κυρία Παρβάνοβα σίγουρα θα γνωρίζει ότι αν φτάσει ένα ασθενοφόρο 5-10 λεπτά νωρίτερα από ό,τι έχει φτάσει μπορεί να έχει σωθεί μια ζωή παραπάνω. Αν βέβαια δεν έχει τις αισθήσει του οδηγός και δεν είναι σε θέση να κάνει τίποτα, κάποιος θα έρθει, θα μας βρει αν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Κάποιος άλλος δηλαδή. Πάντως ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το λάβει η υπόψη της στα πλαίσια και τις οδηγίες για τις οικουμενικές υπηρεσίες. Ωραία. Οι σκιώδεις, οι συγητές, εντάξει. Δύο λεπτά όμως τώρα. Να ακούσουμε τον κύριο Ρίκη από την Επιτροπή. Για να σας ακούσουμε όλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στους εισηγητές και για τη δουλειά τους και για την επιμονή τους. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή αρχή η ηλεκτρονική κλίση. Το αν γίνει όμως υποχρεωτική αλλάζει εντελώ η φύση της. Γιατί αρχίζει και δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Κάποια από αυτά τα ακούσαμε. Το ένα πρόβλημα είναι ότι αν είναι υποχρεωτική αυτή η ρύθμιση, τότε θα πρέπει τα δίκτυα, τα διάφορα κέντρα να προσαρμοστούν. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει γενική εφαρμογή. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το θέμα των κέντρων ε, κλήσης αλλάζει η φύση τους. Γιατί αν τώρα έχουμε ένα εκατομμύριο οχήματα που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα και μετά γίνει υποχρεωτικό το σύστημα αυτό, καταλαβαίνετε πόσες κλήσεις θα δέχεται το κέντρο αυτό. Τα μισά, πρέπει να ξέρετε, μισές κλήσεις είναι κλήσεις όπου δεν ακούγεται τίποτα Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επανοργάνωση ήδη. Αν είναι υποχρεωτικό το σύστημα και οι κατασκευαστές ε, οχημάτων υποχρεωθούν να το προσφέρουν, θα γίνεται τεχνικά, θα γίνεται, δεν υπάρχει αμφιβολία, οικονομικά όμως θα στοιχήσει. Άκουσα τον πρόεδρο να λέει ότι μα πρέπει κανείς αν δεν θέλει να φαίνεται το που βρίσκεται θα πρέπει να μπορεί να αδρανοποιεί το σύστημα αυτό. Υπάρχουν προβλήματα, ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο οπότε δεν θα συνεχίσω για πολύ, αλλά σας λέω, η αρχή είναι πάρα πολύ καλή, αλλά αν γίνει υποχρεωτικό τότε δημιουργούνται χιλιάδες προβλήματα. Αυτό είναι για μένα το ζήτημα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριος Μπακτ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Το... Όλοι συμφωνούμε στους στόχους αυτού του e-call και δεδομένου ότι έχουν αναφερθεί με οργανωτικά προβλήματα, το 80% των οδηγών πιστεύω θα ωφεληθούν από αυτό το δίκτυο, από αυτό το, την κλίση, τον αριθμό ε, δεν προσπαθούμε εμείς να εφεύρουμε τον τροχό, αλλά θέλουμε να εδραιώσουμε κάτι το οποίο τεχνολογικά είναι εφικτό. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει κοινή βούληση. Γιατί η, ο τομέας, ε, ο κατασκευαστικός, ο βιομηχανικός τομέας ακολουθεί διαφορετικό δρόμο από ό,τι η πολιτική βούληση. Εγώ πιστεύω ότι ο τομέας θέλει να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό ως εμπορικό σύστημα και θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτούς που ε, χρησιμοποιούν τον αριθμό αυτό ως πελάτες. Ε, δεν θέλουμε όμως εμείς να συμπαρασυρθούμε σε αυτό τον ε, ε, δρόμο, τον απατηλό δρόμο, διότι βασικά αυτό που δεν θέλουν είναι στις στατιστικές να εμφανίζονται τα, τα στοιχεία τους, για στα ατυχήματα δηλαδή, στα αυτοκίνητα, μάρκες αυτοκινήτων κλπ. Εμείς έχουμε την πολιτική βούληση και θέλουμε να ωφελήσουμε τους οδηγούς, τους πολίτες και γι' αυτό ο συνάδελφός μου Κόχο και η κυρία Σιναλόβα, Σέστατε ε, το ερώτημα και στην Κομισιόν. Ε, μα τι προβλέπει η Κομισιόν εδώ να κάνει. Έχουμε τόσο καιρό συζητήσει το θέμα. Και συμφώνω και με τις φήμες που ακούγονται μάλλον ε, για την Κομισιόν ότι υπάρχουν αντικρώμενες απόψεις μέσα στην Κομισιόν. Να μας ξεκαθαρίσει λοιπόν τη θέση της η Κομισιόν. Η κυρία Φώστερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Συμπρόεδρε. θα επαναλάβω μερικά από αυτά τα θέματα τα οποία εσήγησαν. Ε, πιστεύω ότι η ιδέα αυτή είναι τόσο προσφυλής σε μας ε, και την υποστηρίζουμε όλοι. Εάν το αριθμό είναι 1-1-2, πολύ ωραία και ε, η προσέγγιση είναι πολύ σωστή. Όμως υπάρχουν προκλήσεις όπως τις έχουν υπογραμμίσει άλλα μέλη. Παραδείγματο χάρη, η υπερχρεωτική τοποθέτηση, τοποθέτηση ενός ανιχνευτικού μηχανήματος, στο, ε, μηχανήματος ηλεκτρονικού που θα με εντοπίζει στο αυτοκίνητό μου, θα με ανιχνεύει. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Προτιμώ λοιπόν κάθε προσέγγιση να είναι σε λούσια και όχι υποχρεωτική. Αν θέλει κάποιο να αγοράσει αυτό το, ε, το μηχανηματάκι ανίχνευση θα το πάρει, αλλά όχι υποχρεωτικά. Εν συνεχεία βεβαίως ε, αυτή η κάρτα την οποία θα αγοράζεις κλίσεων βεβαίως όσο πιο πολλές μονάδες αγοράζεις τόσο πιο πολύ θα κοστίζει άρα είναι οικονομικό και το θέμα. Και το τρίτο είναι υποδομή, αναγκαία υποδομή η οποία θα χρειάζεται Εάν κάποιος ζει σε απομακρυσμένη περιοχή υπάρχουν προβλήματα πρόσβαση στο δίκτυο, υποδομής λοιπόν. Επίσης το θέμα της, ε, ε, του, του airbag, της σακούλας ασφαλείας η οποία εκτινάσεται όταν έχει ατύχημα. Πολλές φορές εκτινάσεται χωρίς να υπάρξει ατύχημα, άρα λοιπόν στατιστικά στοιχεία. δεδομένα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές προκλήσεις που απαιτούν πολλές απαντήσεις και Ευχαριστώ όλους για την δουλειά που έκαναν και τους δύο εισηγητές και η συζήτησή μας θα είναι καρποφόρη με βέβαιο. Ο κύριος Higgins, ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα σχόλια των δύο εισηγητών όσον αφορά την καθυστέρηση της Κομισιόν και επίσης τα σχόλια του Μάλκομ Χάρμπορ και της κυρίας Γκούρμε. Είπε ότι περίπου 40.000 άνθρωποι σκοτώνται στους δρόμους μας στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία... Μία... Α, επίσης ο κύριος Κόχο, ο οποίος είπε πρέπει να κάνουμε μία μελέτη σκοπιμότητας κόστους ωφέλους. Μα δεν μπορούμε να ε, ποσοτικοποιήσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Κάθε φορά που ένα αυτοκίνητο βγαίνει από το δρόμο του έχουμε μία ε, χρυσή ευκαιρία μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ας πούμε μία ώρα να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή χρονικο διαστημα α όχι να περιμένουμε μέχρι την επόμενη το πρωί, εφόσον μπορούμε να καλέσουμε αυτό τον αριθμό για βοήθεια. Τώρα, ποιος θα περίμενε πριν από μερικά χρόνια ότι θα έχουμε αυτά τα μηχανήματα GPS τα οποία μπορούν, ε, ε, ε, πλοήγησης τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας εντοπίσουν. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα διαλειτουργικότητος σε μια διασυνοριακή Ευρώπη ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί και πέραν των συνόρων μιας χώρας, δηλαδή θα είναι υπεραδαφικό. Όλα αυτά τεχνολογικά γίνονται. Αν υπάρχει βούληση υπάρχει και το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε ο κύριος Γκρός, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να μην ε, επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν. Εγώ πιστεύω ότι ο στόχος είναι καλός, ο δρόμος προς την επίτευξη δύσκολος. Ε, όταν ψάχνει κανείς για προσκόμματα πάντοτε θα τα βρίσκει. Εγώ προέρχομαι από περιοχή κοντά στα σύνορα και με τις Σαμπίνες ζούμε σε απόσταση 8 χιλιόμετρων. Εάν θέλει κάποιο να επικοινωνήσει με την οδική βοήθεια σε εμά, πρέπει να περάσει από ένα τηλεφωνικό κέντρο. Άρα λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι στη γενική υπηρεσία που θέλουμε να εδραιώσουμε εδώ το 112, προϋποθέτει μία εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδιώκουμε πάντοτε την εφαρμογή νέων τεχνολογιών χωρίς να κοιτάμε από δίπλα τι κάνει το γειτονικό μας κράτος. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε μια ενιαία τεχνολογία. Η τεχνολογία στο Βέλγιο μπορεί να χωρέσει σε ένα μικρό κουτάκι που λέει πού βρίσκομαι, πόσο γρήγορα πηγαίνω, αν υπάρχει καμία συμφόρηση στο δρόμο, τι συμβαίνει, κανένα ατύχημα κλπ. Και μπορεί καμιά φορά να μιλήσω και με τους φίλους μου στο τηλέφωνο. Η τεχνολογία υπάρχει, η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει, αλλά και πάλι σκοντάφτουμε τα ε, διασυνοριακά ε, ε, προσκόμματα, στις, στις, στις, τα εμπόδια τα οποία τυχόν θα συναντήσουμε όταν περάσουμε τα σύνορα. Στις τηλεπικοινωνίες, παραδείγματος χαρή. Ε, καμία φορά το, ε, βγαίνω έξω από το δίκτυο, δεν υπάρχει καθόλου δίκτυο στο τηλέφωνό μου σε 10-15 χιλιόμετρα σε ορισμένε περιοχές, δεν καλύπτεται. Ε, αν λοιπόν θέλουμε αυτό το σύστημα να γίνει υποχρεωτικό, να κοιτάξουμε σαφέστατα ποιοι πρέπει να λειτουργούν αυτό, τον αριθμό, πρέπει να είναι το προσωπικό, το έμπειρο του 112 και οι αρμόδιοι λοιπόν του 112 να λειτουργούν το σύστημα και επίσης να είναι διαλειτουργικό. Μην ξεχνάτε και το γλωσσικό. Πέραν της ε, ε, υπερσυνοριακής ε, τεχνολογίας υπάρχει και το γλωσσικό. Ο συνάδελφός μου από την Ολλανδία που ζει κοντά στα σύνορα επικοινωνεί, καλύπτεται όμως από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της γειτονική χώρας, ας πούμε, της Γερμανίας, άλλη γλώσσα. Λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε ε, και αν τα λύσουμε οι πολίτες μας θα είναι ευγνώμονες. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε για εμπόδια, να, να ψάχνουμε για λύσεις. Ευχαριστώ κύριε Γκρός, λέει ο πρόεδρος. Α, σύμφωνα Πιστεύω ότι δεν συμφωνείτε με μηχανήματα εντοπισμού ραντά της τροχέας για υπέρβαση ταχύτητος. Όχι, όχι πρόεδρε, καθόλου. Απλώς ε, αυτό που διαπίστωσε σήμερα είναι όπως ο Χριστός ότι μπορούμε να μεταμορφώσουμε το νερό σε κρασί, άμα θέλουμε. Απολύτως λέει ο πρόεδρος. Πολύ σωστά. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, μπορείτε κι εσείς να μετατρέψετε σε δύο λεπτά το νερό σε κρασί. Λοιπόν, λέει η κυρία Λίχτεμπεργκερ, έχω και εγώ σοβαρέ επιφυλάξει. όσον αφορά τα δεδομένα, προστασία δεδομένων. Δεύτερον, όταν λέμε ότι οι λύσει για τα δεδομένα θα είναι να, κλείνει κανείς το μηχάνημα, τότε προκύπτουν θέματα τεχνικής ασφάλειας. Άμα το βγάλουμε εκτός λειτουργίας για να προστατεύσουμε τα δεδομένα, αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί. Βεβαίω, προληπτικά θα λειτουργήσουν οι διατάξει ότι κάποιος που έχει αυτό το σύστημα e-call θα έχει το όφελος χαμηλή ταρήφα, ε, χαμηλού κόστους. Τώρα, σε περιοχές ε, δύσκολης πρόσβασης τι θα γίνει τεχνολογικά. Ε, ε, τι θα γίνει σε περιοχές όπου το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει 100%. Τώρα, αν κάποιο βασίζει τα επιχειρήματα στον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων και νομίζει ότι με το e-call αυτομάτως θα λυθεί το πρόβλημα των 40.000 τροχαίων θυμάτων, κάνει λάθο, διότι Εάν κάποιος, ας πούμε, οδηγεί και ε, ε, κατά λάθο ή ε, επίτηδες έχει κλείσει το μηχάνημα για να μην εντοπιστεί στον αυτοκινητόδρομο, τώρα θα, έχουμε, θα έχει αυτομάτως πρόβλημα η ασφαλιστική εταιρεία με την ασφάλισή του εάν συμβεί κάτι. Και με το 112 θα έχουμε προβλήματα και με την παρεμβολή σε άλλα δίκτυα, παραδείγματος χάρη ασθενοφόρων, ή ελικοπτέρων ε, νοσοκομιακών μεταφορών αέρος και επίσης με λανθασμένες κλήσεις ή με κλήσεις φάρσα. Λοιπόν, και αυτά είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βερνιό, Μπερναντέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε παρακολούθησα ως είπε συνάδελφο για την προστασία των δεδομένων και για το γεγονό ότι το 112 θα έχει και αυτά τα όρια του. Όμω, για να θυμίσω όσο είπε και η Data και όσο είπε ο δεν θυμάμαι το όνομά του δίπλα στην κυριολεκτική, εγώ κάθε φορά ξαφνιάζομαι όταν μιλάμε για τη σχέση κόστους-οφελίας. Χέγγιν, Higgins. Όταν ε, μιλάμε για το σχέση κόστου ωφελίας σε περίπτωση που πραγματευόμαστε ανθρώπινες ζωές. Δεν είμαι ιδιαίτερο αυταρχική, ούτε απαιτώ διαρκώς την ε, δεσμευτική υλοποίηση. Όμως κάποιες φορές οι πολίτες έχουν ανάγκη να τους σώζουμε και από τους εαυτούς τους. Ναι προστασία των δεδομένων είναι ένα ζήτημα που το εντάξει, το κατανοώ. Όμω, την ίδια συζήτηση κάναμε και στην Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και εδώ μιλάω ε, υπό την ε, αιγίδα του Προέδρου Μάλκομ, γιατί είδαμε το θέμα αυτό το 2009 με τη σχετική έκθεση, για το 112. Όταν εξετάσαμε το 112, ε, όπου ήμουν υπεύθυνη ε, της έκθεσης. Μίλησα με όλους τους διασώστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μου είπαν ότι μπορούμε να σώσουμε 4.000 ζωές στην Ευρωπαϊκή Υπηρώ μαζί με τραυματίες. Σκεφτείτε και το κόστος, το νοσοκομιακό, της υγειονομικής περίθαλψης. Εδώ μιλάμε για θέματα όπου αναζητούμε την οικονομία, την εξοικονόμηση δηλαδή κονδυλίων. Σκεφτείτε για την υγεία, για τις ανθρώπινες ζωές. Είναι ένα προηγούμενο καθοριστική σημασίας. Και βεβαίω πρέπει να δοθεί έμφαση στι υπηρεσίε 112. Όλε αυτέ οι υποδομέ να συνδυαστούν. Το συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι ανοιχτή σε αυτό το διάλογο και στι προτάσει δηλαδή του Ευρωκοινοβουλίου, είτε για το e-call για τα οχήματα, είτε για το 112. Και σε κάποιο βαθμό βλέπω ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση στα κράτη μιλώ γνωρίζοντας πολύ καλά τα της χώρας μου. Δεν είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία και την περασμένη εβδομάδα είδα μια τεράστια αφίσα ε, κοντά στο σπίτι μου που λέει σε περίπτωση επίγουσα ανάγκη. Ε, καλέστε το 17 για την πυροσβεστική, το 12 για την αστυνομία. Ε, μα τι να πω, δεν έχουμε πολιτική βούληση στην Ευρώπη για να εξυπηρετήσουμε όσους ζουν στο έδαφος μας. Να το πούμε καθαρά είναι θέμα κόστου, απλώ είναι θέμα πολιτική βούληση. Για το θέμα λοιπόν του e-call και σε συνδυασμό και για το 112. Μιλήσαμε για τους σχεδιαστές των οχημάτων και τους εκπροσώπους των αυτοκινητοβιομηχανιών. Το είπε η συνάδελφος. Κάποια, όπως το πεζοπασάτε, έχουν ήδη εξοπλιστεί τα αυτοκίνητα με το σύστημα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει εμπορική αξία, εμπορικό όφελος και για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Τώρα να μην είναι υποχρεωτικό σε αυτοκίνητα και να προσπαθήσουμε τα μικρότερα οχήματα ή μέσων κυβικών να μην έχουν αυξημένο κόστο, απαγορευτικό για κατηγορίε πολιτών να τα αγοράσουν, εντάξει. Όμω εδώ, από την άποψη της πολιτική βούλησης, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει πραγματικά να στραφεί στα κατημέλη και να το πει στου υπουργού τη κάθε μια μα χώρα. Έχουμε σημαντικέ αποφάσει να λάβουμε για σκοπούς ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και γιατί μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την προστασία της καθημερινής ε, ζωής και της ίδιας της ζωής των πολιτών. Εάν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, σε περίοδους κρίσης όπου η Ευρώπη απορρίπτεται διότι είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για όλα τα κρατικά προβλήματα, πρέπει τέτοια θέματα να τα προωθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δισταγμού. Να συζητήσουμε με όλους τους υπευθύνου ε, του ντοσχέ αυτού και να προχωρήσουμε, κάνοντας έκκληση και στα κάτι μέλη. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τρεις εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση MOVE, IMSO και Θα δώσω δύο λεπτά στον καθένα σας κυρίες και κύριοι, και κυρία, μάλλον. Θα ξεκινήσω από τον ε, κύριο, με τον κύριο Και επίσης η βασική ερώτηση, πολύ διπλωματικά, ε, γιατί καθυστέρησατε τόσο, κύριε Γκονζάλη. <clears throat> Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ευχαριστήσω όλο το Κοινοβούλιο για αυτή την έκθεση, που έχει κερδίσει τη συμπάθειά μα όχι μόνο σήμερα, αλλά όλα τα τελευταία χρόνια μέσω τη πρωτοβουλία για το e Να πω ότι συμφωνώ μαζί σα σω χρονοτριβήσαμε για την ενσωμάτωση του e στα οχήματα. Όχι γιατί δεν γνωρίζουμε τα ωφέλη του e αλλά γιατί επεξεργαζόμαστε το θέμα, όπω είπατε, από το 2002. Και το επεξεργαζόμαστε α, επί τη θελούσια βάση. Είδαμε ότι στην αγορά δεν λειτουργεί στην πράξη το σύστημα. Πολύ λίγα οχήματα έχουν εξοπλιστεί με αντιστάσει των καταμελών. Δοκιμάσαμε πάντα την εθελούσια μέθοδο και πραγματικά καθυστερεί ιδιαίτερω. Γι' αυτό λοιπόν πλέον επιμένουμε για τα δεσμευτικά μέτρα. Για το θέμα της προστασίας δεδομένων να κάτι. Για το e που προωθούμε δεν σημαίνει ότι ο καθένας που θα οδηγεί το όχημα θα μπορεί να ανοιχνεύεται. Το 112 δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Δεν είναι κανείς συνεχώς συνδεδεμένο στο δίκτυο. Μόνο σε περίπτωση ατυχήματος. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι υπέρμαχοι του συστήματος αυτού. Αποφασίσαμε ότι η ηλεκτρονική κλίση πρέπει να προωθηθεί και ο σχεδιασμός, ο ηλεκτρονικός σχεδιασμός να σέβεται και τα ιδιωτικού βίου. Έπειτα υπήρξαν πολλά, πολλές παρατηρήσεις για το βαθμό υλοποίησης από την επικοινωνία, τη σχετική επικοινωνία της Επιτροπής. Ξέρετε ότι προτείνουμε κάποια ρυθμιστικά μέτρα. Ο συνάδελφος από τις Γενικές Διευθύνσεις ε, Enterprise και MOVE θα τα θυμίσει αυτά. Όμως όσα ανακοίνωσε η Επίτροπος κρού τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν στόχος υλοποίησης το 2015. Θα συνεργαστούμε λοιπόν ώστε να αναβαθμιστεί και το κομμάτι της κατασκευής αυτών των οχημάτων και το τηλεπικοινωνιακό και της υποδομής. Τώρα έχουμε σταθεί στο θέμα των τηλεπικοινωνιών. Έχουμε σχετικέ συστάσει, βλέπουμε τι εκθέσει των 100 μελών και βλέπουμε τι γίνεται με του παροχή ε, υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Δεν θέλουν να υπάρξει και μεταχείριση των διαφορών δικτύων μεταξύ του και στηρίζουν το 112. Όμω πρέπει όλε τι εκθέσει να τι μελετήσουμε προσεκτικά. Εάν ε, κάτι μα ξεφύγει, θα φροντίσουμε να το συμπληρώσουμε μέσα από τι εκθέσει και τι παρατηρήσει των 100 μελών. Έπειτα τεχνικά ζητήματα που ετέθηκαν έχουμε διεξοδικότατη μελέτη αντικτύπου. Περάσαμε πολλούς μήνες βλέποντας την σχέση κόστος ωφελίας και υπάρχουν πολλοί αριθμοί που αφορούν το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος του οίκων. Αποτιμούμε λοιπόν τώρα την εκθέση αντικτύπου. Βλέπουμε τον αριθμό ατυχημάτων και υπάρχουν πολλά ατυχήματα στις στους επαρχιακούς δρόμους όπου καθυστερεί η παροχή υπερκουσών υπηρεσιών. Στη Φιλανδία έγινε μια σχετική μελέτη και ε, φάνηκε ότι από την καθυστέρηση των επιγόντων περιστατικών να τα αποκριθούν ε, χάσαμε πολλέ ζωέ. Πολλέ θα είχαν χαθεί. Αυτό μα δείχνει μελέτη αντικτύπου. Τώρα προ το κόστο, ε, αποτιμήσαμε το κόστο και τι ενδεχόμενε ωφέλη και βλέπουμε ότι τα ωφέλη, άσχετα από τη συζήτηση για το πώς θα αξιολογηθεί το κόστος της ανθρώπινης ζωής ή τα τραύματα ή εναπηρίες, τα ωφέλη είναι περισσότερα από το κόστος. Είναι σαφές. Εάν με ρωτάτε τώρα ποια είναι τα διαφορετικά κόστη για τα οχήματα περιλαμβάνοντα τη μελέτη αντικτύπου σχετική αριθμή, Ξέρουμε πόσο θα πανηρώθανε το κάθε στοιχείο, αλλά στα οχήματα, εφόσον ενσωματωθεί το σύστημα αυτό, μειώνεται το κόστος ήταν πάρα πολλέ όμω ερωτήσει, δεν μπορώ να τα ανακεφαλαιώσω όλα. Ε, δύο λεπτά μου δώσατε, α συμπληρώσουν οι συνάδελφοι. Το κόστο. 15 ευρώ. Για τη μελέτη δικτύπου υπολογίσαμε 150 ευρώ θεωρητικά και πάλι είναι μεγαλύτερο τα ωφέλη. Για την υποδομή και για τον ε, Τσέχο συνάδελφο, εάν εξοπλιστεί σωστά, αν εξοπλιστεί σωστά η υποδομή του 112 είναι περιθωριακό το κόστος. Αλλά εξαρτάται από το ποιον φορέα θα καταστήσουμε υπεύθυνο να λαμβάνει τις κλήσεις του 112 ή κάποια άλλο αριθμό και το κόστος δεν θα ξεπεράσει τα εκατοντάδες ή κάποιες χιλιάδες ευρώ. Πάντως το θέμα είναι να υπάρξει φωνητική σύνδεση, ε, ελάχιστα δεδομένα και κάποια χρήση της τακτικής ε, που ήδη χρησιμοποιείται στα 112. Πρέπει εδώ να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες, να περιορίσουμε δηλαδή τον ρυθμό κλήσεων. Ε, ήδη εδώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Πρέπει και η ομάδα δράσης για το e να τοποθετηθεί εδώ, γιατί λύσεις υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν ήταν ε, τεχνολογικώ ουδέτερη, γι' αυτό ζητούμε από τους οργανισμούς τυποποίηση να μας δώσουν τεχνολογικές λύσεις με ανοιχτά πρότυπα για τεχνολογικούς σκοπούς. Σας ε, αφήνω το λόγο αφού ολοκλήρωσα, νομίζω ότι μακρηγόρησα ήθελα να αποστείλω ένα συγκεκριμένο μήνυμα στην Επιτροπή. Όλοι θα μιλήσετε ή ο καθένα ξεχωριστά, διότι πρέπει να ε, περιορίσετε το χρόνο σα. Τέλο πάντων, η απάντηση ήταν όλοι θέλουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, μην εξαντλήσετε την πρόσβαση την υπομονή μου. Κυρία Ντέρνερ από τη Γενική Διεύθυνση μου. Ευχαριστώ. Α, έχω δώσει, έχω σπρώξει ένα μέρος της ομιλίας μου στον ε, επικεφαλής της ΙΜΣΚΟ. Το e-call 112 ήταν πάντοτε μια πρωτοβουλία την οποία καλύπτει η Κομισιόν και στο πρόγραμμά μας το 2012 περιλαμβάνεται όπως τονίστηκε στην προηγούμενη έκθεση από του, του Κοινοβουλίου του κυρίου Κόχο και θέλω να πω ότι έχουμε θέσει τις προδιαγραφές για το PSEP, e για την κλίση εκτακτής ανάγκης, το μηχάνημα κλπ. Και υπάρχει στην, στο κεφάλαιο 8 της, του σχέδιου γνωμοδοτήσεως και η Κομισιόν επεξεργάζεται αυτές τις προδιαγραφές ε, και θα τις μεταφέρει σε μια κατεξουσιοδότηση πράξη πριν από το τέλος του χρόνου αφού εξεταστεί από την ομάδα πυρογνωμόνων. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, όταν κάποιος ανέφερε delegated κατεξουσιοδότηση πράξη είδα μερικά απορριμμένα βλέμματα. Η κυρία Μπόνι φυσούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Απλώ να συμπληρώσω για το τεχνικό σκέλο του συστήματο. ECOL. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει μια, ένα σχέδιο πρόταση για να δούμε το νομικό πλαίσιο για τα οχήματα κατηγορία M1, όπω τα εμπορικά οχήματα. Οι λεπτομέρειε οι τεχνικέ αυτή τη στιγμή ε, ολοκληρώνοντα την εξέτασή του από τι αρμόδιε υπηρεσίε τη Επιτροπή, λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω τι διάφορε επιλογέ με τα ωφέλη του. Πρέπει να τονίσουμε ότι για τα οχήματα θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το σύστημα όταν τα των τεχνικών προδιαγραφών τηλεπικοινωνιών και οδικής ασφάλειας έχουν εξεταστεί πλήρως μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει να επιβληθούν οι υποχρεώσεις για το νέο σύστημα. Σας ευχαριστώ. Οι συγητές, δεν είμαι βέβαιος αν καταλάβαμε ποιος είναι ο καθήλυν υπεύθυνο εδώ με τόσα παρεμβάσει από του βουλευτέ. Η κυρία Συναλόβα όμω να ξεκινήσει και μετά ο κύριο Κόχ. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, ειλικρινά, για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, που αναμφίβολα θα εμπλουτίσουν την έκθεση αυτή επανερχόμαστε, τουλάχιστον πολλές από τις ερωτήσεις σας ε, επανέρχονται στην ιδέα του κατά πόσο πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή σε θελοντική βάση το σύστημα ηλεκτρονικής κλήσης. Είναι κάτι που συζητάμε εδώ και πολλά κλείνουν οι απόψεις. Συμφωνώ με όσα ακούστηκαν εδώ, ότι δηλαδή είναι θέμα πολιτικής βούλησης το κατά πόσο θέλουμε ή όχι να προσανατολιστούμε ε, σε αυτή τη βάση. Οι τεχνικές λύσεις ή όλα τα τεχνικά ζητήματα λύνονται στην περίπτωση που αποφασίσουμε ότι το θέλουμε. Θέλω να αντιδράσω λίγο σε κάποιες παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με το κόστος. Πώς να υπολογίσουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής, πώς να υπολογίσουμε με τι κόστος, τι ζωές που μπορούμε να κερδίσουμε από την ηλεκτρονική κλίση. Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί και όχι το οικονομικό κόστος. Ευχαριστώ πάντως για τις παρατηρήσεις σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε πολλά ερωτήματα. Για την περίπτωση των κλήσεων που δεν είναι πραγματικές, εδώ πρέπει να δούμε τις άστοχες. Εδώ πρέπει να δούμε πότε μπαίνει σε δράση το σύστημα ανάλογα με το τύπο του ατυχήματος και αν δεν μπορεί να υπάρξει φωνητική επαφή να μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για τη σοβαρότητα του ατυχήματος από διάφορα άλλα στοιχεία, από άλλους δείκτες που θα περνάνε στο σύστημα. Πάντως τα ΠΕΣ και ΑΠΕ πρέπει να ε, αναλύονται από τα κέντρα υποδοχής των κλήσεων. Εκείνοι πρέπει να καταλαβαίνουν κατά πόσο πρόκειται για ηλεκτρονική κλήση όχι έπειτα το πώς ε, θα παρακολουθούν τα οχήματα, το είπα και στην αρχή. Αυτό το σύστημα παρακολούθησης θα μπαίνει σε εφαρμογή μόνο από τη στιγμή που γίνεται ατύχημα. Δεν παρακολουθεί δηλαδή το σύστημα το όχημα καθόλου τη διάρκεια της πορείας του, μόνο από τη στιγμή που γίνεται ατύχημα. Ε, έπειτα υπάρχει και το θέμα της ουδετερότητας ε, τεχνικά. Μα το κείμενο λέει ε, ναι, τεχνολογικά ουδέτερο, αλλά σεβόμενη τις προδιαγραφές ασφάλειας. Είναι προφανές ότι μία κινητή εγκατάσταση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από το ίδιο το ατύχημα. Για το θέμα των υποδομών, του Κέντρου Υποδοχής των Κλήσεων, το 112 δηλαδή, και εδώ έχουμε πει ότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία πρέπει να φροντίσουν για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Ευχαριστώ πάντως που υπενθυμίσατε και την οδηγία για τις οικονομικές ε, υπηρεσίες. Όντως είναι ευθύνη των κρατών μελών οι οικουμενικές υπηρεσίες. Ο συνάδελφος θα συμπληρώσει φαντάζομαι. Ναι, πολύ σύντομε παρατηρήσεις. Επειδή δεν μου απάντησε η Κομισιόν στο βασικό μου ερώτημα, εάν ισχύει αυτό που ο κύριο Ταλιάνη, δηλαδή το μορατόριο μου. Δηλαδή καμία ρύθμιση για την αυτοκινητοβιομηχανία με ενδιαφέρει, με καίει αυτό. Βεβαίω, δεν μπορούμε να αποφύγουμε όλα τα ατυχήματα. Όμως η χρυσή αυτή ώρα, η κρίσιμη μετά το ατύχημα, μπορεί να σώσει πολλέ ζωέ. Δεύτερον, οι υπηρεσίες ε, άμεσης ε, ανάγκης διάσωσης είναι, είναι σημαντικές ε, να λειτουργήσουν σωστά, να έχουν το, σωστό δίκτυο κλήσεων Ιδίω σε θέματα, σε ατυχήματα που γίνονται από πεθυσμένου οδηγού. Ούτε ένδο δεν θα έπρεπε να σημειώνεται, αλλά δυστυχώ γίνονται και εάν υπάρχει ανάγκη μέσω της επίγουσας κλήσης πρέπει να πάνε οι διασώστες, οι σωστικές υπηρεσίες. Ποιος θα πληρώσει, πρέπει όλοι να συνυπογράψουν ένα μνημόνιο ε, συνεννόησης, ένα memorandum of understanding για να γίνει σωστή κατανομή του κόστους. Δεν είναι και τόσο τεράστια, τεράστιες οι δαπάνες πρέπει να φροντίσουμε μια τέτοια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί ακόμα και αν κοστίζει κάτι στο κράτος μέλος. Εν συνεχεία, το ότι ε, ε, κάποιος θα μας παρακολουθεί συνέχεια, το αόρατος κατάσκοπος θα μας παρακολουθεί συνέχεια. Δεν είναι σωστό αυτό, διότι το σύστημα αυτό δεν θα λειτουργεί ε, και δεν θα μας παρακολουθεί συνέχεια. Αλλά όταν θα λειτουργεί και θα μας εντοπίσει και θα το χρειαστούμε, θα είμαστε ευγνώμονες. Η κοινή βούληση, εντάξει, πρέπει να υπάρχει αλλά ποιο ήρθε πρώτα, η κότα ή το αυγό. Η αυτοκινητοβιομηχανία λέει, αν δεν λειτουργήσει το σύστημα στα κράτη-μέλη, δεν χρειάζεται να το τοποθετήσουμε στα αυτοκίνητα. Τα κράτη-μέλη λένε ότι αν δεν τοποθετηθεί το μηχάνημα από τι αυτοκινητοβιομηχανίε, δεν χρειάζεται να εδραιώσουμε το σύστημα. Η κότα και το αυγό λοιπόν. Τώρα το κόστος των κατασκευαστών, το είπαμε, βασικά είναι θέμα λογισμικού, software. Δηλαδή, όχι τεράστια δαπάνη, τόσο τεράστια δαπάνη. Και τέλος, εάν περιμένουμε έως ότου κάθε δυνατό πρόβλημα ή πιθανό πρόβλημα έχει λυθεί μέχρι ότου εισαχθεί αυτό, αυτή η υπηρεσία θα έχουμε περάσει το 2012 και το 2112. Λοιπόν, ε, πρέπει το ταχύτερο να δημιουργήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το σύστημα και να λειτουργήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσά και όλους τους σκιώδες εισηγητές και όλους όσοι πήραν το λόγο στη συζήτηση αυτή. Η προθεσμοί για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 8η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Πρόθεσή μας είναι η επόμενη κοινή συνάντηση, τη προσκλήση της ΣΥΜΚΟ, να γίνει την Τετάρτη 30 Μαΐου. 11 με 12 και 30 τότε θα εξετάσουμε και τις τροπολογίες που θα έχουν υποβληθεί. Προθεσμία λοιπόν 12 το μεσημέρι της 8 Μαΐου και επόμενη ε, κοινή μας συνεδρίαση 30 Μαΐου την προσκλήση της ΙΜΚΟ για να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Μάρκο, υπάρχει μήπω κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ και που προεδρεύσατε τόσο καλά τη συνεδρίαση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ και 30 Μαΐου θα έρθουμε εμείς σε εσάς. Συνεπώς, αυτή η συγκεκριμένη συνεδρίαση λύγει έτσι, αλλά οι συνάδελφοι από την Επιτροπή των Μεταφορών να μείνουν εδώ γιατί έχουμε τις εκθέσεις του κυρίου Κράμερ. Εντάξει, Μάικλ, η σειρά σου. Okay, if people are... Uh, ε, καθίστε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ναι, Όποιος θέλει να κουβεντιάσει, μπορεί βέβαια, αλλά εκτός αθούσης παρακαλώ. So if people are moving... Λοιπόν, Βγείτε όσοι θέλετε. Ένα λεπτάκι, Μιχάλη, περίμενε να εγκαταλείψουν την αίθουσα όσοι φεύγουν και μετά. There three Έχουμε τρεις γνωμοδοτήσεις του κυρίου Κράμερ όσον αφορά τη διαθετική πολιτική Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μάκλη. Ευχαριστώ. Είναι δύο ε, ε, γνωμοδοτήσεις είναι για ε, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κατάργηση του Κανονισμού, ειδικέ διατάξει για με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και εν συνεχεία το Ταμείο Συνοχή. Είχαμε την τελευταία φορά ακούσει ένα πολύ ωραίο κάτι που είχε πει ο Τσόρτσιλ χρειαζόμαστε μια στρατηγική, αλλά πού και πού, πού και πού χρειαζόμαστε και αποτελέσματα. Θαυμάσια ρίση λοιπόν αυτή του Τσόρτσιλ που ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε στρατηγική αλλά λείπουν τα αποτελέσματα. Διότι στα διαστρωτικά ταμεία έχουν προβλεφθεί από το 2014 μέχρι το 2020 180 εκατομμύρια ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πάλι ένα τεράστιο ποσό και μια χρηματοδότηση 85, μέχρι 85%. 31 δισεκατομμύρια υπάρχει, θα διατεθούν σε σχέση με τη, τη Euro Facility, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διευκόλυνσης και αυτά τα ταμεία έφρα και το Ταμείο Συνοχής δηλαδή το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη και το Ταμείο συνοχή θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουμε ή όχι. Εμένα ο στόχος μας είναι ε, να συνδυάσουμε τις ε, επενδύσεις αυτές των υποδομών με την ε, πολιτική του, μέχρι το 2020 και τα προγράμματα Natura και άλλα που εμπίπτουν στα διαφορετικά ταμεία. Γι' αυτό πρέπει η στρατηγική μας να βασίζεται στην αηφορία και στην αποτελεσματικότητα. Ορισμένα παραδείγματα. Όλα τα ε, σχέδια, τα προγράμματα της εσωτερικής ναυσιπλοείας και η διεύρυνση του ποταμού Έλβα ε, σκοντάφτουν στις, στα παράλληλα προγράμματα ε, ανάπτυξης των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων. Μέχρι τώρα μόνο 11 από 27 εσωτερικά λιμάνια έχουν χαρακτηριστεί ως ε, αποτελεσματικά. Δηλαδή ότι η χρηματοδότηση ας πούμε θα είναι αποδοτική και θα έχει αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα... Ε, 15, 16 λιμάνια έχουν χαρακτηριστεί ως μη ωφέλιμα, μη αποτελεσματικά. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ πού θα επενδύουμε τα χρήματα στις κατάλληλες, στους κατάλληλους αποδέκτες και όχι πόσα χρήματα και συνέχεια να ζητάμε. Τώρα έχουμε ένα τούνελ από την Βιέννη που θα βοηθήσει να υπάρχει έξοδος προς την Αδριατική ε, μέσω των... Ε, Μέσω του τούνελ αυτού θα διευκολυνθεί πάρα πολύ η πρόσβαση από τις βόρειες χώρες μέσω Βιέννη στην Αδριατική και επίσης θα δημιουργηθούν και περιολές θέσεις εργασίας κατά τη δημιουργία της σύραγγας αυτής. Επίσης, ε, η διασύνδεση Erfurt-Nirenbergi. Εκεί ε, διεπιλέχθηκε ένας ε, δρόμος, χαράχτηκε ένας δρόμος με πάρα πολλά τούνελ και με πάρα πολλές γέφυρες. Λίγο πιο νότια να είχε χαραχθεί ο αυτοκινητόδρομος θα ήταν πιο φτηνά, πιο σύντομα και πιο αποδοτικός ο δρόμος αυτός και θα, είχαμε εξοικονομήσει δισεκατομμύρια τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα αν κοιτάξουμε γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι συγκεκριμένα παραδείγματα. Εδώ και 30 χρόνια έχουμε η στρατηγική, αλλά, αλλά έχουμε ακόμα μία κουρελού μπαλωμάτο, δηλαδή ένα, μία μπαλωματική στρατηγική σε στυλ κουρελούς που δεν μπορούμε να, τη να την συνδυάσουμε, που δεν μπορούμε να την συγκεράσουμε, που δεν μπορούμε να την υλοποιήσουμε διασυνοριακά, διότι σκοντάφτουμε στον, ε, στους εθνικούς σοφινισμούς. Μέχρι τώρα το ε, Ταμείο Περιφοριακής Ανάπτυξης χρηματοδοτούσε 60% αυτοκίνητο, 20% σιδηρόδρομους, ένα ελάχιστο ποσοστό ποδηλατόδρομους κλπ. Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας τώρα για τις μεταφορές. Πρέπει να προσαρμόσουμε τους στόχους μας με τις μελλοντικέ ανάγκες. Το Ρότερνταμ, παραδείγματο χάρη, είναι ο μεγαλύτερος διάδρομος για την αυσιπλοεία και κάθε κάθε 2-3 λεπτά φτάνει ένα μεγάλο τρένο με ένα σειρμός δηλαδή με προϊόντα για το λιμάνι. Έχουμε όμως προβλέψει στο διάδρομο Καλσουρού η Βασιλεία μόνο 180 εκατομμύρια και 3 δισεκατομμύρια Ούλμ Στουτγάρδη, μια διαδρομή δηλαδή η οποία δεν έχει καμία σχέση και κανένα όφελος ε, για τις ε, ε, μεταφορές εμπορευμάτων θα χρηματοδοτεί με 3 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς λόγο. Ε, θέλουμε να προωθήσουμε την, τις περιφερειακές ε, μεταφορές ε, και, να, και ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις περιβαλλοντικές ανάγκες μειώνοντας τους ρήπους από τα καυσέρια. Ξέρουμε ότι ο Υπουργός Μεταφορών Ράμζαρος στη Γερμανία είπε ότι 90% των οδηγών ε, ε, ε, κυκλοφορούν, διανύουν λιγότερο από 6 χιλιόμετρα κάθε φορά που μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Κατά μέσο όρο 90%. Δεν είναι αυτό σωστό, γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να συνδυάσουμε την αηφορία στις οδικές μεταφορές με τις χαμηλές εκπομπές ρήπων και το σεβασμό στις περιβαλλοντικές ανάγκες και να προσέξουμε να μην ξοδεύονται, να μην δαπανώνται λανθασμένα κονδύλια. Ακόμα και στις ανεπτυγμένες περιοχές πρέπει να προσέξουμε. Η Κομισιόν έγραψε να μην δώσουμε δεκάρα, δεκάρα στις ανεπτυγμένες περιοχές για τις ε, μεταφορές. Μα άμα δεν δώσουμε μια δεκάρα, επειδή είναι ανεπτυγμένες οι περιοχές, πώς θα μειώσουμε τις, εκπομπέ τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε την αρχή της αηφόρεως ανάπτυξης, θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέψουμε και πιστώσεις για τις ανεπτυγμένες περιοχές, για τη μείωση των ρήπων. Ε, ε, αηφόρος τουρισμός, και αυτόν πρέπει να τον προωθήσουμε. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας ο τουρισμός. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός μπορεί να βλάψει, μπορεί να καταστρέψει, αλλά ένας σωστός τουρισμός μπορεί να οδηγήσει σε αηφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος τα παραρτήματα είχαν επιπλέον δείκτες και θέλουμε να συμπεριλάβουμε, να τους συμπεριλάβουμε. Παραδείγματο χάρη τον αριθμό των διασυνοριακών συνδέσεων, τον, ε, ε, η σχέση των, ε, των στοιχείων εκπομπής διοξιδίων με τουριστικές μεταφορές. Ας πω ένα παράδειγμα. Το 1972 Γερμανία με Πολωνία είχε 18 συνδρομικές γραμμές καθημερινές καθημερινές. Μετά από 32 ε, χρόνια υπάρχουν μόνο 10, 10 σειρμοί που πηγαίνουν μεταξύ Γερμανία και, Γερμανίας και Πολωνίας. Είναι τρελό, αλλά είναι πραγματικότητα. Εφόσον δηλώνουμε ότι το μεταφορικό μας δίκτυο είναι ευρωπαϊκό, και ο άξονας Βαλτικής Αδριατικής λένε ότι θα κοστίσει πάρα πολύ και θα αρπάξει πάρα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, επιτρέπουμε ταυτόχρονα τη μείωση σιδηροδρομικών μεταφορών και γραμμών οι οποίοι πραγματικά ήταν ωφέλιμοι. ορισμένες τροπολογίες που έχω συντάξει. Θα τις αλλάξω διότι θέλω να καλύψω ορισμένες ιδέες μελών μας, παραδείγματο χάρη όχι αποφυγή αλλά ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους, εκεί συμφωνώ. Επίσης συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, όχι λόγω της στρατηγικής αλλά λόγω των, της έλλειψης αποτελεσμάτων και επίσης θέλουμε ιδέες για να ενισχύσουμε το ρόλο των νέων κρατών μελών όπου σημειώνονται και τα μεγαλύτερα ελλείμματα. Ε, περιμένω με μεγάλη ε, ανυπομονησία την περαιτέρω εργασία μας τις τροπολογίες και η προθεσμία τροπολογιών είναι 7 Μαΐου. 7 Μαΐου. Ε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω να σημειώσω τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Κράμερ για την εργασία του και την, ε, τις επικοδομητικές συζητήσεις που έχουμε ήδη κάνει και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι αυτά τα ντοσιέ είναι σωστά δεδομένου ότι στο όλο θέμα της χρηματοδότησης των μεταφορών είχαμε ζητήσει 16 δις, μας δώσαν 8, όταν στην περιφερειακή ανάπτυξη δόθηκα 40. Άρα λοιπόν αυτός ο τομέας μεταφορικής κινητικότητας είναι πολύ σημαντικός. Θέλω όμως και κάτι να αλλάξω από αυτά που είπε ε, του Churchill. Εγώ θα πω ότι χρειαζόμαστε την πράσινη πολιτική, η στρατηγική αν θέλετε, αλλά που και που να αλλάζουμε και κέντρο βάρους και άλλα κέντρα βάρους. Ε, τα, το Ταμείο Συνοχής ε, και τα διορθωτικά κονδύλια, αν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε όπως προτείνει η Κομισιόν, πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μας προς αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο εδώ, αλλά να σεβαστούμε ακριβώς ε, τη χρήση αυτής της έννοιας της συνοχής όπως ε, την προτείνει η Κομισιόν στην πρώτη έκθεση είμαι εγώ ε, σκιώδης εισηγητής, αλλά στη δεύτερη έκθεση, τροπολογία 2 επί του άρθρου 8, αναφέρονται οι περιφέρειες και λέει ότι εκεί όπου υπάρχουν ε, ε, είναι ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν θα πρέπει να πληνθούν περιττέρω κονδύλια. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε για να μην διαγράψουμε την μεταφορική κινητικότητα. Τώρα, να αποφύγουμε τελείως το εξωτερικό κόστος στο μέλλον, αυτό πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο για μένα, διότι είναι υπερβολικά περιοριστικό. Να αποφύγουμε, ναι, αλλά όχι να εξαλείψουμε τελείως, να αποφύγουμε, ναι, να μειώσουμε, να αμβλύνουμε το εξωτερικό κόστος, ναι. Όπως επίσης η βιοπικιλία, η βιοπικιλότητα. Ε, πολλές φορές παρουσιάζεται αυτό ως ε, δικαιολογία, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι για τη βιοπικιλότητα, δεν χρειάζεται να την προβάλλουμε τόσο στεναρά. Πιστεύω ότι πάντοτε μπορούμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση ε, και αυτά τα θέματα, αυτές τις επικεφαλίδες αν θέλετε, πρέπει να τις χρησιμοποιούμε με σύνεση. Επίσης θα ήθελα να μου μια διευκρίνηση για την τροπολογία 29 όπου αναφέρεσαι στην ανάγκη ψηλότερης χρηματοδότησης. Εάν κατάλαβα εγώ καλά, βάσει της, της γαλλικής στρατηγικής θα κάνω έναν αυτοκινητόδρομο, θα έχω καλά έσοδα, προβλέπω ε, καλά, καλές προσόδους ας πούμε, αλλά πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό χρηματοδότησης, Έτσι έχει. Ε, έτσι είναι, αυτή είναι η σωστή ιδέα. Ε, δεν έχω καμία άλλη παρατήρηση. Ελπίζω να, ε, να συνεργαστούμε σωστά και να καταλήξουμε σε συνεργαστικές τροπολογίες. Eh, κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ. Ε, και ευχαριστώ και τον κύριο Κράμερ για τις προσπάθειες που έχει κάνει ώστε να μας εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια την επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι όπως έχει η κατάσταση και με τις δυσκολίες που έχουμε με το Συμβούλιο που μάθαμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η μάχη θα είναι πολύ σκληρή. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε κάτι καλύτερο. Πιστεύω πάντως ότι εκτός από τις λεπτομέρειες χρειαζόμαστε και μια άλλη πολιτική. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ριζοσπαστικοί σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για το ΦΕΝΤΕΡ. Δεν θα υποστηρίξει επενδύσεις ή υποδομές στις πιο αναπτυγμένες περιοχές. Μα ξέρουμε ότι είναι βασικό η πολιτική συνοχή στα διορθωτικά ταμεία χρησιμεύουν για να βοηθούν τα κράτη-μέλη ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες περιοχές υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι θύλακες με μεγάλες ανισότητες, με προβλήματα ανταγωνιστικότητας, ανισορροπία δηλαδή ανάμεσα στο κέντρο μιας πόλης και την περιφέρεια ή ανάμεσα στο βουνό και την πεδιάδα δίπλα. Μέσα ακόμα δηλαδή και στην ίδια περιοχή. Το να λέμε ε, ανεπτυγμένη περιοχή οπότε δεν δίνουμε τίποτα, όχι δεν με βρίσκει σύμφωνη. Και να ξέρετε ότι από τις πολλές περικοπές οι επικεφαλείς κάποιων περιφερειών αναπτυγμένων έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν μπορούν πια να καλύψουν τους κατοίκους εκεί. Μπορεί το 2008 να έστεκε. Σήμερα πάντως όχι πείτε μου μια τέτοια αναπτυγμένη περιοχή για να σας πω πού υπάρχουν τα προβλήματα μέσα σε αυτήν την ε, θέμενη ανάπτυξη ή τέλος πάντων την ανάπτυξη που φαίνεται αλλά που δεν υπάρχει παντού σε αυτή την περιφέρεια. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον αποκλεισμό αυτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κράμερ για το τρόπο που χειρίζεται το όλο το σχέδιο για την προσέγγιση που έχει καθορίσει. Και για το έργο του νομίζω θετικό είναι το γεγονός ότι πλαισιώνοντας το θέμα του ζήτησε και προτείνει στην Επιτροπή Μεταφορών να εντάξουμε το όλο θέμα και στην προοπτική του 2020. Όλο ο προγραμματισμό μα πρέπει να υπόκειται ακριβώ και σε αυτή τη σκοπιά. Για να μην έχουμε διαρκώ νέα φάση προγραμματισμού. Και για να παραθέσω κατά λόγια κάποιο μαζί με την καλή βούληση και τα καλά αποτελέσματα που ανέφερε και ο Τσέρτσιλ, το σημαντικό με τη στρατηγική είναι να υπάρχει μία στρατηγική. Δεν μπορεί να προσαρμόζεται η στρατηγική κάθε φορά που υπάρχει μια διασταύρωση με κάποιο άλλο ζήτημα. Οι προοπτικές άλλοτε είναι πιο άνετες και άλλοτε πιο σφιχτές. Πρέπει λοιπόν να πω ότι είναι θετική αυτή η τοποθέτηση. Επίσης, για την τροπολογία 25, μια μικρή αρνητική παρατήρηση, ζητάτε να προβλεφθεί δημοσιονομική γραμμή ξεχωριστή στους κρατικού προπολογισμού για τους ποδηλατοδρόμου και τους πεζοδρόμους. Εδώ μάλλον συγκεκριμένο προγραμματισμό χρειαζόμαστε και δεν το βρίσκω σωστό αυτό ως γενική ένδειξη. Επίσης για την τροπολογία 28, ο όγκος των επενδύσεων για τους ποδηλατοδρόμους, εδώ θα μπορούσαμε να μιλάμε για, για όγκο των βιο, της βιώσιμης ευθυούς κινητικότητας, χωρίς να περάσουμε σε τόσο συγκεκριμένες αναφορές. Όμως βρισκόμαστε σε φάση προπαρασκευαστική ούτως ή άλλως του όλου, της όλης συζήτησης, γι' αυτό θα παραμείνω και εγώ σε τέτοιο πνεύμα. Τώρα, μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό του συγκεκριμένα. 10 δις υπέρ της διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη. Αυτά τα διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προορίζονται στις περιφέρειες που έχουν πρόσβαση στα Ταμεία Συνοχής. Όμως να μην ξεχνάμε και το εξής. Η κεντρική αυτού χαρακτήρα διαχείριση κεντρική μάλλον κεντρικού χαρακτήρα διαχείριση, μπορεί να έχει επιπτώσεις αρνητικές σε περιοχές με ελλείμματα διοικητικά, ε, προγραμματισμού. Εδώ λοιπόν το κριτήριο όποιος ε, φτάσει πρώτος είναι και εκείνος που θα εξυπηρετηθεί θέτει σε δυσχερή θέση τις ε, περιοχές που ούτω ή άλλω αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τελευταία λοιπόν παρατήρηση, πολύ θετική, εκτιμώ και στηρίζω πλήρω το λίμα του τουρισμού μεταξύ των κοινών δικτών και την εισαγωγή του λίματος του τουρισμού μεταξύ των κοινών δικτών. Αυτό είναι σημαντικό και για σκοπούς οικονομικής ανάπτυξης που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι από τα αναπόσπαστα στοιχεία των σκοπών ενός τομέα όπως των μεταφορών. Κύριε Ζήλε. Ευχαριστώ. Πρέπει εδώ να πω ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Κράμερ οδεύει στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που θα ήθελα να σχολιάσω σε άλλη φάση, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ μας, όπως η έμφαση των ε, επενδύσεων, οι διώσιμες μεταφορές μέσω του Ταμείου Συνοχής. Ναι, πολύ καλή προσέγγιση αυτή. Και με την αιτιολόγηση που υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση. Ο μηχανισμός για τη διασύνδεση της Ευρώπης ε, προβλέπει 10 δις ευρώ όμω να μην ξεχνάμε τα προβλήματα των χωρών που με 2,2% του ΑΕΠ δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του Ταμείου Συνοχή. Για κάποια κρατή μέλη, λοιπόν, δεν θα υπάρχει στήριξη από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που ξεπερνά το στενό πλαίσιο της πολιτικής μεταφορών. Τώρα για συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρόταση 5 με ικανοποιεί ιδιαιτέρως, διότι ο Μίκαελ δίνει μεγάλη έμφαση στην πτώση του σιδηρού παραπετάσματος ή για τη διασύνδεση Δύσης και Ανατολής. Εδώ δεν υπάρχουν οι απαραίτητε υποδομές, Καλά λοιπόν κάνετε και δίνετε έμφαση στο σημείο αυτό. Για την 8 τροπολογία, εκεί που προτείνεται μια κατανομή των ποσών μεταξύ μεγίστων και ελαχίστων για τους σιδηροδρόμους, τους πεζοδρόμους και τους ποδηλατοδρόμους. Εδώ έχω κάποιους ενδιασμούς σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. μπορεί να υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης στους δρόμους εφόσον εμείς θέσουμε κατόφλια στα ποσά που θα δαπανηθούν. Εάν δεν υπάρξει οδικό σύστημα λόγου χάρη, πώς θα υπάρξουν ποδηλατόδρομοι στη συνέχεια. Πώς θα κυκλοφορεί ο κόσμος για να φτάσει στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Ποια θα είναι τα σημεία διασύνδεσης για την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν κάποιε αποκλήσει απόψεων, αλλά είμαι ευνοϊκά διακειμένο προ την ε, συνολικά. Ε, ε, ε, ευχαριστώ και εγώ. Και ευχαριστώ τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για την ε, παρουσίασή του, αλλά και για τη συνεργασία του με τους σκιώδες εισηγητές. Και συμφωνώ μαζί του για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βασιστεί περισσότερο στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020 και στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, όπως επίσης και στις αρχές αλληλεγγύης και μείωση των διαφορών ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Αυτά είναι οι στόχοι της πολιτικής συνοχής εξάλλου. Συμφωνώ και με τον εισηγητή για το ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε και να κινητοποιήσουμε νέους τρόπους κινητικότητας βιώσιμη κινητικότητας. Τα μαζικά μέσα μεταφοράς, για παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι κατά προτερότητα επιλογή των πολιτών. Τώρα, για τις αδυναμίες και πώς αυτές θα παληθούν μέσω της αναθεώρησης των δικτύων. Ο εισηγητής εδώ υπογραμμίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που πρέπει να είναι ο ρόλος της επιλογής των προγραμμάτων. Ζητάω λοιπόν και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα σύνολο δικτών, μετρήσιμων δικτών, που να μας επιτρέπει να απαλείψουμε τις παρεξηγήσεις. Ο εισηγητή επίση υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα ενίσχυση των ελέγχων εξάντε και των προτέρων. Σωστά, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε και στα προγράμματα ποιότητας, αλλά και τους ελέγχους εξ μετά. Υπογραμμίζω και εγώ το θέμα του τουρισμού. Σίγουρα πρέπει να του δώσουμε περισσότερη σημασία. Όσον αφορά τις τροπολογίες τώρα του εισηγητή που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό κόστος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ ίσως θα έπρεπε να μου εξηγήσει περισσότερο τι ακριβώς εννοεί, σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεται. Δυστυχώς δεν συμφωνώ και με τον ορισμό του συγκεκριμένου ποσοστού για τα διάφορα είδη μεταφορών. Τροπολογία 8. Διαφωνώ επίσης και με την τροπολογία 29 που έχει να κάνει με τους γενικούς κανόνες όπου θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα προγράμματα από τα οποία έχουμε σαφές κέρδος. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, δεδομένων των στόχων της συνοχής. Και θέλω να υπογραμμίσω επίσης και την ανάγκη να μην ξεχνάμε τον κύριο στόχο της πολιτικής συνοχής που είναι η εξισορρόπηση των υποδομών μεταφορών σε όλες τις περιφέρειες, άρα και στις λιγότερο αναπτυγμένες. Αυτό μην το ξεχνάμε. Για τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου πάντως θα τα ξανασυζητήσουμε έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ο κύριος Ραπκάρη. Ευχαριστώ. Η έκθεση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης έχει ως στόχο να προωθήσει επενδύσεις που θα ενισχύσουν και την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο κύριος Κράμερ στη, ε, στην τροπολογία του 2015 αναφέρεται σε ένα διαλειτουργικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό σιδηροδρομικό δίκτυο που θα υποστηρίζει ε, το πολυσχηδές ευρωπαϊκό μεταφορικό δίκτυο μέσω επενδύσεων. Μέχρι εδώ καλά. Όταν άκουσα στο γραφείο μου αυτά που έλεγε ο κύριος Κράμερ, ε, κάπως εξεπλάγει όταν άκουσα ότι υπάρχει ο διάδρομος Βαλτικής Αδριατικής μέσω της Αυστρίας. Ε, βέβαια η Αυστρία βρίσκεται σε αυτό το διάδρομο και ε, δεν είναι δυνατόν άμα δεν σκάψεις τούνελ και άλλα έργα υποδομής να υλοποιηθεί αυτός ο βαλτικο-αδριατικός διάδρομος από το Ελσίνκι δηλαδή, μέσω των γνωστών κρατών, μέσω των Άλπαιων και τα λοιπά που να φτάσει στα βόρεια αδριατικά λιμάνια, σαφώς θα παρουσιάσει μια προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία στην ανάπτυξη. Και γι' αυτό εξεπλάγει τον άκουσα τα σχόλιά σας ότι δίνονται τόσα κονδύλια για αυτό το διάδρομο και δεν δίνονται αλλού που είναι πιο χρήσιμα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να καταλάβετε ότι για να γίνει αυτός ο μεταφορικός διάδρομος χρειάζονται τεράστιες ε, επενδύσεις έργων και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ ε, ωφέλιμο και προς την κατεύθυνση των κοινών μας στόχων. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξετε θερμότατα ε, το έργο αυτό και βεβαίως το συνεπαγόμενο κόστος και όχι να το επικρίνετε, διότι θα είναι ένα έργο το οποίο θα αποδειχθεί λίγα αναποτελεσματικό. Ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Α, έχω. Έχω, έχω. Ευχαριστώ πρόεδρε οι τροπολογίες που προτάθηκαν από τον κύριο Κράμερ και αναφέρονται στο άρθρο 5 ε, πρέπει να θα πρέπει εκεί να προσθέσουμε δύο ξεχωριστές παραγράφους που θα λένε που θα παραπέμπουν στην πρόταση της Κομισιόν. Υποστηρίζω την αστική ανάπτυξη και την διάθεση 5% των κονδυλίων σε αστικά προγράμματα, σε προγράμματα αστικών περιοχών. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Υπήρχε μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο δύο βαθμίδων, διάφορες προσεγγίσεις, διάφορες απόψεις και το, το πρόγραμμα σύνδεσης της Ευρώπης πρέπει να γίνει πιο σαφές στο, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Διότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των δύο ταμείων όσον αφορά τις ε, αιτήσει για επενδύσεις. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εάν στις ανεπτυγμένες περιοχές θα δώσουμε ή θα δεν θα δώσουμε αναπτυξιακά κονδύλια, αναπτυξιακές πιστώσεις. Euh, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πνεύμα διαλεκτικότητας που έδειξε σε όλες τις συζητήσεις. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι όταν, όταν μιλάμε για ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης, μιλάμε για περισσότερο από 90% χρηματοδότησης για τις μεταφορές. Ξανά ευχαριστώ λοιπόν το webstream και τον κύριο Κράμερ που ακούει τόσο καλά και τα δικά μας σχόλια και εμείς τον ακούμε. Τέλος παντών, από την πολυετή χρηματοδότηση, το 90% ε, αφορά τα περιφερειακά ταμεία. Λοιπόν, έχει τεράστιο δημοσιονομικό βάρος αυτό. Επίσης, ο σκιώδης εισηγητής για τα ταμεία συνοχής, να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ταμεία αυτά και στηρίζω τον εισηγητή στις τροπολογίες που επισημαίνουν την αναπερκή πρόοδο, το πόσο δρόμο έχουμε ακόμη να κάνουμε για τους στόχους του 2020 και τους περιβαλλοντικούς στόχους και για την έμφαση που δίνει στον τουρισμό. Τώρα για το ποσοστό διακριτικής μεταχείρισης και επιλογής για ορισμένο τύπου προγράμματα δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα αυτό γιατί σε κάποια από τα ταμεία ορισμένα δις έχουν να μεταφερθεί μέσω της διευκόλυνσης προς ε, την ε, διαδικασία αυτή διασύνδεσης ή οδοί και οι δρόμοι αποκλείονται τελείω. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να μα απασχολήσει. Από το να προβλέψουμε και το δικό σύστημα ένα μηχανισμό διακριτική μεταχείρισης θα προκαλέσει εξέγερση. Και θα βλάψει και του στόχου διασύνδεση που θέλουμε να πετύχουμε. Θα υποβάλουμε λοιπόν κάποιε τροπολογίε ώστε να επικεντρωθούμε στην βοήθεια που θα έχει και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αλλά και εδώ νομίζω ότι λίγο πολύ συμφωνούμε. Τώρα, για τα αποτελέσματα που διώκουμε και την μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μεταξύ των οριζόντιων προτεραιοτήτων μας, ιδίως με το σύστημα ευφυών μεταφορών, έναν άλλο τρόπο να προσθέσουμε αξία ευρωπαϊκή στα ταμεία συνοχής, χρειάζεται και τεχνική συνδρομή και προτάσεις για τους δείκτες. Τώρα για το ΦΕΝΤΕΡ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μία μόνον παρατήρηση. Υπάρχει μια τροπολογία το γνωρίζει η κυρία Γιάλα νομίζω, που θέλει να, να θέσει ένα ανώτατο όριο στην χρηματοδότηση του Φεντερ. Τα ταμεία συνοχής με 30 δις από τον προπολογισμό για τις μεταφορές κατά ουσιαστικά ανταποκρίνονται σε 40% στα περιφερειακά ταμεία. Αυτό ισοδυναμεί. Δηλαδή, εάν πάρουμε αυτά τα 30 ε, από αυτό το ταμείο, θα, θα εξαλείψουμε άλλα 40. πώς θα γίνει η διασύνδεση της Ευρώπης και πώς ε, με την προηγούμενη υπηρεσία που υπήρχε τα 20 δις μας ενδιαφέρουν θα τα διασώσουμε. Λοιπόν, από τα κονδύλια χρηματοδότηση των μεταφορών θα χάσουμε τουλάχιστον 20 δι ε, με τον τρόπο αυτό. Να προσέξουμε λοιπόν πολύ με την πρόταση αυτή και να απορρίψουμε την ε, δυνατότητα αποκλεισμού των μεταφορών. Να μην ξεχνάμε ότι η κρίση έχει, πλήξει και τις ε, χώρες που παραδοσιακά είχαν καλή ανταγωνιστικότητα, τώρα γίνονται όλο και πλέον ελληματικές. Ε, η περικοπή από τη χρηματοδότηση των περιφερειακών ταμείων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις μεταφορές. Και θα ήταν θανατηφόρε αυτή τη στιγμή τέτοιου είδου ε, δεσμεύσει για τον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ λοιπόν την προσοχή των συναδέλφων. Εάν τα πράγματα τα αφήσουμε ω έχουν ω προ την ανταγωνιστικότητα, θα είχαμε σεισμό στην χρηματοδότηση των μεταφορών. Θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά δεν θα μας επιτρέψει η διευκόλυνση Connecting Europe να αντισταθμίσουμε αυτό το σεισμό. Από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μπέρκοβιτς. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και υψηλής ποιότητας. Πολλά από όσα συμπεριλαμβάνει εκεί ευθυγραμμίζονται και με τα όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Στρατηγική 2020. Από πλευράς της Επιτροπής λοιπόν έχουμε κάποια σχόλια προκειμένου να υπάρχει κάποια ισορροπία. Θα σας τα πω αυτά. Στην πρότασή μας προσπαθήσαμε κατά πολύ να συμπεριλάβουμε τις κλιματικές αλλαγές και σε ολόκληρο το πρόγραμμα και με ορισμό στρατηγικής, και με διάφορους παράγοντες στα προγράμματα αυτά καθε αυτά, αλλά και στο πρόγραμμα επιλογής δραστηριοτήτων επιτόπου. Γι' αυτό, ενώ καταλαβαίνουμε βέβαια πολύ καλά τις ανησυχίες σας, πιστεύουμε ότι καλύπτονται. Ιδιαίτερα ε, μέσω της αρχής ορυπαίνων πληρώνει. Οπότε το θέμα δεν είναι τόσο πολύ θέμα προθέσεων, είναι πιο πολύ θέμα διατύπωσης. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα, το θέμα της ισορροπίας. Μία από τις προτάσεις και στους τρεις και στα τρία θέματα έχει να κάνει με το πώς θα συμπεριλάβουμε τις μεταφορές στην οικονομία χαμηλού άνθρακα. Εδώ όμως αυτό είναι πολύ περιοριστικό δεδομένο των στόχων της συνθήκης για τις μεταφορές. Πάλι πρέπει να σας πω ότι συμμεριζόμαστε πολλές από τις ιδέες σας. Για παράδειγμα βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα σας σύνδεση με το 2050 και το χαμηλό άνθρακα αλλά ίσως μερικές φορές ο τρόπος με τον οποίο το κάνετε οδηγεί σε επιπλέον διοικητικό άχθος και μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να πετύχουμε συνένεση. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι διαχειριστικές αρχές και οι διάφοροι αρμόδιοι να συμφωνήσουν. Ένα άλλο θέμα, που είναι πάλι θέμα διατύπωσης, έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό ε, αναφορών σε δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Όσα αναφέρεται μπορούν να χρηματοδοτηθούν, εντάξει μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις με ε, το focus, να ένα παράδειγμα. Πάντως ένας μεγάλος κατάλογος, κυρίως αν δούμε τις τροπολογίες άλλων επιτροπών, δεν βοηθούν, γιατί έτσι η προσοχή του κόσμου στρέφεται από τους στόχους μας σε άλλα πράγματα. Τώρα θέλω να έρθω κάπως σύντομα στη χρηματοδότηση των υποδομών στις πιο πλούσιες περιφέρειες, κάτι το οποίο αναφέρθηκε. Εντάξει, μπορεί να δίστανται οι απόψεις εδώ, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι λέει η πρόταση της Επιτροπής. Λέει ότι δεν θέλουμε να, να χρηματοδοτούμε βασικές υποδομές. Δηλαδή υψηλή κλίμακα. Τι είναι αυτό για μας, είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι υψηλή ταχύτητας ε, δρομικέ γραμμές τι πλώσιε περιφέρειες, που είναι πάνω από το 90% του μέσου όρου της ε, Ένωσης. Γιατί προτείνει νέα κατηγορία μεταβατικών περιοχών η Επιτροπή. Και γιατί το κάναμε αυτό, όχι γιατί πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι οι πόροι που διατίθεται για τις πιο πλούσιες περιοχές είναι πολύ χαμηλή. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πιο μικρά προγράμματα, μικρότερης κλίμακας, μπορεί να είναι μια προστιθέμενη αξία. Βέβαια, οι χώρες μέλη που επιλέγονται για το Ταμείο Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτηθούν ανεξάρτητα από το τύπο του προγράμματος. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια μικρή εξαίρεση που έχει να κάνει με τους διαθέσιμους πόρους. Κάτι τελευταίο τώρα για τον τουρισμό. Για μας ο τουρισμός, και προσπαθώ να σας εξηγήσω γιατί το παρουσιάζουμε έτσι, ε, είναι γιατί για μας ο τουρισμός είναι πολύ σημαντική η οικονομική δραστηριότητα. Δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεισφέρει μέσω των στόχων ε, του 2020 να συνεισφέρει λοιπόν στη δημιουργία ανάπτυξη, θέσεων απασχόληση και προστασία του περιβάλλοντο. Γι' αυτό εμεί δεν θέλουμε να βάλουμε τον ε, τουρισμό να το συνδέσουμε με ένα μόνο συγκεκριμένο τομέα. Για του δείκτε που μα ζητήσαν, εντάξει, να κοιτάξουμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε του δείκτε. Και ευχαριστώ να συζητήσουμε με τον εισηγητή περισσότερο σε λεπτομέρειε για αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Πολύ Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για να απαντήσω. Μα πρόκειται για βασικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τις μεταφορές και τα εφή δίκτυα. Νομίζω ότι είναι κακό μήνυμα αυτό που στέλνετε, γιατί για μια μικρή συγχρηματοδότηση τελικά δεν έχουν κίνητρο οι περιοχές αυτές. Είναι ένα κακό, στραβό μήνυμα, αρνητικό. Τη στιγμή που πρόκειται για βασικές υπηρεσίες για τους ε, πολίτες. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να στέλνουμε ένα τέτοιο μήνυμα, ακριβώ επειδή είναι μικρός ο προπολογισμό. Για μένα είναι προτεραιότητες όχι μόνο των πιο πλούσιων περιφερειών, αλλά της Ευρώπης προτεραιότητες. Ο Μάικλ. Αλλά και αυτό το θέμα, ε, γιατί αυτό με δυσκολεύει και εμένα. Αυτό το θέμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Αυτό με ενδιαφέρει. Μια γραμμή υψηλής ταχύτητας μπορεί να ξεκινάει σε μια πλούσια περιφέρεια ή να καταλήγει σε μια πλούσια περιφέρεια, περνάει όμως και από άλλες. Έτσι κι αλλιώ, σε μια συνδρομική γραμμή έχουμε δύο άκρες. Έτσι το βλέπω εγώ την τελευταία φορά. Ναι, εντάξει, εκτός αν είναι κυκλική γραμμή και πάμε γύρω-γύρω. Μάικλ, εσύ τώρα. Ναι, μπορώ να σας πω το παράδειγμα, ένα παράδειγμα. Νιρεμβέργη Έρφουρτ χρηματοδοτήθηκε αυτή η διαδρομή και συνεχίζει προς το Μέναχο. Αλλά από το Μόναχο στο Ζάλτσπουργκ δεν υπάρχει ούτε καν η ιδέα επέκτασης, αλλά ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη διοχετευθεί ε, από τον αυτοκίνη, στον αυτοκινητόδρομο Ερφούρτη ε, προς Μόναχο ας πούμε. Αλλά τη συνοριακή περιοχή από από Ζάλσμπουργκ ε, δεν την έχουμε αφήσει απ' έξω, ούτε καν τη σκεφτήκαμε. Διότι ε, δεν υπήρχε ούτε η βούληση ούτε τα κίνητρα τα κατάλληλα να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση ώστε να περάσει και τα σύνορα. Τώρα, για τον, αυτά που είπε ο Ματιού Γκρός. Ναι, βεβαίως, σωστά τα είπε. Όταν ε, φτιάξω έναν αυτοκινητόδρομο και μετά βάλω διόδια, έχω έσοδα, εντάξει. Όταν όμως κάνω μια συνδρομική γραμμή, υπάρχουν Τελεί στου συνδρομικού σταθμού, ή άμα περνά τα, τα σύνορα α πούμε. Οπότε χρειάζομαι ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για να περάσω και να φτιάξω τις ε, γραμμές. Δεν μπορούμε λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε διόδια στους σιδηρόδρομους, αλλά μπορούμε να μαζέψουμε έσοδα κάπως διαφορετικά, να μην χρηματοδοτήσουμε τους σιδηρόδρομους, επειδή μπορούμε να βάλουμε διόδια στους αυτοκινητόδρομους και να χαρατσώνουμε τους οδηγούς. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να παραμελήσουμε τα τρένα. Ανάπτυξη περιφερειών και πόλεων. 2,2% είναι η, χρηματοδότηση, η πρόταση χρηματοδότησης της Κομισιόν ε, για χρηματοδότηση περιφερειών. Εάν περιφέρειες έχουν ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2,2% εκπίπτουν από το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Τώρα, στα αστικά κέντρα, στις μεγαλοπόλεις, δεν φτιάχνουν αυτοκινητόδρομους, αλλά φτιάχνουν έναν δρόμο, ας πούμε, βασικό για την πόλη 10 χιλιόμετρων. Εμπίπτει αυτό στα μεγάλα έργα ή δεν εμπίπτει. Από απόψεως μεγέθους δεν εμπίπτει. Από απόψεως όμως περιβαλλοντικού προβλήματος εμπίπτει. Διότι αν τον δρόμο αυτό των 10 χιλιόμετρων το χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Α, και μία παρατήρηση. Walking ε, μεταφράστηκε... Α, το, το, η λέξη walking μεταφράστηκε κάπως διαφορετικά στα γερμανικά, άσχετο με την ουσία. Ε, τώρα, ε, αν τα πάρω τα 3,5 δισεκατομμύρια της συνοχής και μπορώ να τα διαθέσω εκεί που θέλω, θα ήταν πάρα πολύ ωραία στον διάδρομο Βαλτική-Αδριατικής. Όμως υπάρχει και η Τσεχία η οποία συνορεύει και η Τσεχία λέει θέλω και εγώ μερίδιο διότι και οι μεταφορές στη Τσεχία είναι, σημαντικό, είναι σημαντική, σημαντικός τομέας παρόλου παρόλο που η διακίνηση στο Δούναβι έχει συρρυκνωθεί σημαντικότατα τα τελευταία δέκα χρόνια και δεδομένου ότι περνάει από την τυχεία. Οι, οι τα εσωτερικά ποτάμια λοιπόν έχουν συρρυκνωθεί, οι διασυνοριακές μεταφορές στα, πρώην, ανατολικά κράτη έχουν συρρυκνωθεί. Πρέπει λοιπόν πολύ προσεκτικά να δούμε πού θα διαθέσουμε τα κονδύλια, σε ποιους άξονες. Και διαρωτώ με, ε, γιατί αποκλείεται, ε, το, το άλλο ζήτημα που συζητήσαμε, γιατί αποκλείεται τις μεγάλες αστικές περιοχές. Ε, γιατί τις αποκλείει η Κομισιόν. Δεν είναι δυνατόν να αποκλείσουμε τελείως περιοχές που είναι ανεπτυγμένες. Όπως σας είπα υπάρχει περιβαλλοντικό στοιχείο. Εν συνεχεία, ε, εάν επενδύσετε 40% στους σειρμούς, δηλαδή στους σιδηροδρόμους, θα καταφέρετε να κερδίσετε την πλειοψηφία κάποια παρατήρηση γίνεται εκτός μικροφώνου. Δεν, δεν άκουσα. Α, τουλάχιστον 40% για σιδηροδρόμους. Ναι, σωστό. Α, τουλάχιστον 40%. Αλλά μην ξεχνάτε τα νέα κράτη-μέλη. Βουλγαρία, Ρουμανία τα τελευταία 10 χρόνια, τα μία συνοχή και τα κονδύλια που πήρανε. Νομίζω από τα κονδύλια, από τι επενδύσει που πήρανε, 99% πήγανε στου δρόμου και τίποτα σχεδόν στους σιδηροδρόμους. Πού, είναι το 40% λοιπόν. Εγώ πήγα, πήγα σε αυτές τις χώρες με, το τρένο και έχασα και πολλή ώρα, γιατί δεν ήταν καλές οι συγκοινωνίες. Λοιπόν, η Αυστρία θέλει τρία τούνελ να φτιάξει. Θέλει να φτιάξει τρία τούνελ, έτσι, τώρα θέλει να τα φτιάξει περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ λένε οι εμπειρογνώμονες θα κοστίσουν. Αυτά τα τρία τούνελ. Και οι εμπειρογνώμονες λένε ότι η Αυστρία δεν τα έχει αυτά τα λεφτά. Και είναι λάθος της διότι έσπρωξε όλες τις μεταφορές στους δρόμους και όχι στους σιδηρόδρομους. Και ρωτάω τώρα, τι θέλετε, τι είναι καλύτερο, για τον Γκράτ και την Κλάγκενφούρτη είναι ενδιαφέρον ένα τούνελ. Αλλά για την Ευρώπη, από την Πρατισλάβα ας πούμε, είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθούν οι σιδηρόδρομοι. Τι θέλετε επιτέλους. Και στη Γερμανία προβλέπουμε τούνελ. Εγώ είμαι εναντίον αυτών των πολυδάπανων έργων. Ε, άλλη παρατήρηση. Α, μην ξεχνάτε και τα, την πολιτιστική κληρονομιά που προστατεύεται από την UNESCO. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ο κύριος Πικέ. Τι, α, τον κάλυψα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις σας. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε πολύ ωραία και θα καταφέρουμε να συντάξουμε ένα ενδιαφέρον έγγραφο. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 7 Μαΐου το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 31 Μαΐου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο μάλλον. Ιούλιο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι υπό τα διάφορα. Απλώς να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες Δευτέρα 7 Μαΐου. Στις 3. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και τους Γερμανείς. Λήξη τη συνεδρίασης.